Καθίστε παρακαλώ. <laughs> so, Σας παρακαλώ να καθίσετε αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίσατε παρακαλώ για αναλαμβάνει στα αγγλικά ο πρόεδρος και θέλω να καλωσορίσω την ε, καλεσμένοι μας, αλλά ο κύριος ε, Λάινεν ζητάει το λόγο. Παρακαλώ, γιο. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω την ε, Επίτροπό μας. Αλλά πρέπει να πούμε κάτι για την αντιπροσωπεία μας στη διάσκεψη Ρίο συν 20. Θέλετε να το κάνουμε τώρα ή αφού θα έχουμε ακούσει την Επίτροπο. Και εγώ υποστηρίζω τον συνάδελφο Λάινεν και ίσως θα πρέπει να αναφερθούμε τώρα στο θέμα αυτό γιατί και η Κομισιόν εμπλέκεται στο θέμα αυτό. Ε, νομίζω όμως ότι θα πρέπει να δείξουμε σεβασμό προς την ε, κυρία Επίτροπο. Το κάνουμε μετά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ υποστηρίζω την αίτηση του Γιολάινεν να συζητήσουμε ενδεχομένω ακόμα και τώρα το θέμα αυτό. Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν για την απόφαση η οποία ελήφθη σε σχέση με την αντιπροσωπεία μας και ποια είναι τα συμπεράσματα που πρέπει να αντλήσουμε. Ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θέλει να έχει μια θέση μέσα στις ε, διαπραγματεύσεις στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής για τη Γη. Γιατί αυτό φαίνεται να είναι το μήνυμα το οποίο ε, δίνει η απόφαση των συντονιστών σήμερα το πρωί. Μπορούμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Σήμερα το πρωί είχαμε τη συνάντηση των συντονιστών. Είναι σημαντική βέβαια αυτή η διάσκεψη Ρίο συν 20. Ο εισηγητής μας είχε οργανώσει και μια συζήτηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πράγματι προσκαλέσαμε τα Εθνικά Κοινοβούλια εδώ στις Βρυξέλλες και υπήρξε μια μεγάλη συμμετοχή από τη δική τους πλευρά. Και εγώ πάντα έχω αντιληφθεί ότι πάντα είναι καλόδεκτη η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά, διότι είμαστε και νομοθέτες και θα πρέπει και εμείς να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες πλειοψηφίε, να κάνουμε τα απαραίτητα νομοθετήματα για όλα αυτά τα θέματα και επομένω είναι σημαντικός και ο ρόλος μας στη διάσκεψη για το όριο. Είπα στους συντονιστές πώς προβλεπόταν να είναι η πορεία την ε, της συνδιάσκεψης, ποιος ήταν ο προϋπολογισμός μας, έχουν δεκαπλασιαστεί οι τιμές των ξενοδοχείων, έχουν φτάσει στα 1000 ευρώ και επομένως το κόστος θα ανέλθει σε περίπου 20.000 ευρώ ανά Είχαμε να κλείσουμε τα ξεροδοχεία αυτά για μπλοκ εβδομάδων που αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μονάχα κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης αλλά και σε χρονικές στιγμές που δεν θα υπήρχε κανένας εκεί. Και εμείς έχουμε εκφράσει την ε, διαμαρτυρία μας γιατί μας υποχρεώσανε να νοικιάσουμε σε ένα υπόγειο μια αίθουσα συνεδριάσεων για 10.000 ευρώ. Γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα οργανωτική να έχουμε μια άλλη αίθουσα συνεδριάσεων. Εγώ έκανα κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσω ότι θα έχουμε ένα χώρο για να προσκαλέσουμε άλλους κοινοβουλευτικούς και μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και τώρα έχουμε τις εξής δυνατότητες. Να μην πάμε καθόλου. Είναι μια δυνατότητα και αυτή ήταν και η άποψη των άλλων συντονιστών, το μεγαλύτερο, του μεγαλύτερου μέρους των συντονιστών. Η άλλη δυνατότητα θα ήταν να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό μας, να τον ε, ξεπεράσουμε δέκα φορές και να ζητήσουμε μια έγκριση από τη συνέλευση των Προέδρων, αλλά οι οργανωτές μας έθεσαν μια καταληκτική προθεσμία μέχρι τις 5 Μαΐου ώστε να πληρωθούν μέχρι τότε όλα τα ξενοδοχεία και χωρίς την απόφαση της συνέλευσης των Προέδρων δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια υπέρβαση. Και δεν έχουμε πάρει μια έγκριση προς την κατεύθυνση αυτή. Η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων θεώρησαν ότι εμείς δεν θα πρέπει να αποδεχτούμε μια τέτοια κατάσταση και επομένως τέσσερις πολιτικές ομάδες έκαναν την πρόταση ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει μεν να έχει τουλάχιστον τον εισηγητή στο Ρίο για να εκπροσωπηθεί εκεί, ώστε να μεταφέρει τις απόψεις μας όπως αναφέρονται στην έκθεσή μας, όπως έχουν καταγραφεί λοιπόν στο ψήφισμά μας, ότι πρέπει λοιπόν να είναι παρόν τουλάχιστον ο εισηγητής, ο κύριος Γκεμπράντι, και θα είναι ο εισηγητής αυτό αφ' αυτού μία μονομελής ε, αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ λυπηρά φυσικά. Αλλά είχαμε το πρόβλημα με την Οργανωτική Επιτροπή στο, στο Ρίο. Όταν έχει κανείς να καλέσει όλο το πλανήτη ουσιαστικά, τότε μπορεί θαυμάσια να αποφασίσει τι θα κάνει και ποιον θα δεχτεί ή όχι. Αλλά εμεί έχουμε ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τον προπολογισμό μα και την αντίδραση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού όπου εμείς δεν ήμασταν ε, μέσα, μέσα στους φτηνότερους αλλά στους ακριβότερους σε ό,τι αφορά τις ε, αποστολές των αντιπροσωπείων θα φτάναμε στις 200.000 ευρώ σε συνολικό κόστος αυτό πράγματι έχει λυπήσει πολλούς συναδέλφους οι οποίοι θέλαν να είναι παρόντες σε αυτή τη διάσκεψη κορφής. Ήταν μια από τις καλύτερες ευκαιρίες να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία μας έχουν απασχολήσει και ο κύριος Γκεμπράντι, ο οποίος είναι ε, πρόεδρος, αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας και εισηγητής, θα πρέπει εν πάση περιπτώσει, να πάει στο Ρίο για να παρουσιάσει τι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα βιοπικιλότητα, κλιματική αλλαγή κτλ. Λοιπόν, από τη στιγμή που είχαμε συζητήσει τα θέματα αυτά έχουν εκραγεί ουσιαστικά το συνολικό κόστος. Αν θέλετε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. έγινε πρόταση ψηφίσματο. Αυτό το κατάλαβα. Ήμασταν διάφοροι. Ο Καλ Χάις Φλόρες, εγώ, η Κορίν Λεπά, η κυρία Μπελιέ, ο Μιρλόσκαβη, η κυρία Λιωτάρ. Εμείς προτείναμε το ψήφισμα. Φυσικά πρέπει να σκεφτούμε και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, ας μην πάμε. Και α διαμαρτυρηθούμε στη βραζιλιάνικη κυβέρνηση, γιατί επιτρέπει τέτοιε συμπεριφορέ γιατί επιτρέπουν όλα αυτά τα πράγματα. Ή θα πάμε όλοι ή θα πάει κανένα. Ε, ευχαριστώ. Κατόπιν ο Γιώλαν Λάιν. Μετά Κρις Ντέιβις και τα λοιπά. Γιώ. Ε, εντάξει, να μην ξοδεύουμε λεφτά, συμφωνώ, σε... και τόσα πολλά λεφτά για δωμάτια που δεν θα τα αγοράσουμε, έτσι. Αν είναι εκβιασμός λοιπόν ε, των ξενοδόχων του Ρίο, πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Και να στείλουμε ένα μήνυμα και να πούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αυτές τις συνθήκες δεν, θε, δεν έρχεται. Η εναλλακτική είναι, νομίζω το είπε ο Βιτόριο, να στείλουμε μια μικρή αντιπροσωπεία αυτούς ε, που στήριξαν ε, το ψήφισμα, ένας από κάθε ομάδα. Για τα ξενοδοχεία δεν ξέρω τι κάνει η Επιτροπή των Περιφερειών ε, και τα το κλαμπ και τα που θα στείλουν 300 άτομα για τρεις μέρες. Η υπόθεση βρωμάει εδώ πέρα. Εγώ λέω να μην πάμε. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε να πρέπει να κλείσουμε τα δωμάτια για 6 μέρες μήνυμου με 600 ευρώ τη. νύχτας. Αν μπω στον υπολογιστή, εγώ θα βρω για 5 μέρες δωμάτια με πολύ λιγότερα λεφτά. Μάλιστα, επόμενος ομιλητής είναι ο Chris Davis. Απλούστατα κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω τη θέση σας. Αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο. Το ερώτημα είναι αν θα στείλουμε έναν ε, εκπρόσωπο ή κανέναν. Η δυσκολία για μένα είναι πως ε, ο πρόσωπος του Κοινοβουλίου, του Προέδρου, είναι μέλος της ομάδας μου. Εγώ θεωρώ πως πρέπει να στείλουμε τον εκπρόσωπό μας, του Κοινοβουλίου εννοώ, και αν τύχαινε να είναι του ΕΛΚ ε, θα το δεχόμουν. Έτσι. Αν υπήρχε πίεση μάλιστα θα ζητούσα από τον κύριο Γκερμπράντη να αντικατασταθεί από κάποιον του ΕΛΚ. Πρέπει να έχουμε έναν και τα υπόλοιπα να διαμαρτυρηθούμε. Σωστά. Ευχαριστούμε, Chris Davis. Judith Merkis. Πρώτα απ' όλα, λυπούμε για το ότι ακυρώθηκε η αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρά το ότι όντως είναι σκανδαλώδες το ότι τα ξενοδοχεία του Ρίο βρήκαν ε, ευκαιρία με τη Σύνοδο να τα οικονομήσουν. Υποτίθεται ότι είναι για το περιβάλλον, την παγκόσμια κλιματική δικαιοσύνη, την εξάλληψη της φτώχειας, πώς θα χρησιμοποιούμε τους πόρους μας. Η Βραζιλία ξέρει να χρησιμοποιεί τους πόρους της και ελπίζω να ωφελήσει το σκοπό αυτό. Αλλά συμφωνώ με τους συναδέλφους. Ή όλοι ή κανένας. Ή συμφωνώ με τον Chris Davis πως ε, το κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπηθεί. Αλλά έχουμε ήδη δύο εκπροσώπους. Ε, ο ένας είναι ο εκπρόσωπος ε, του Προέδρου και ο άλλος ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μας. Και νομίζω πως σε καιρούς λιτότητας το να εξοδεύουμε τέτοια ποσά για αυτή την αποστολή είναι σκανδαλώδες. Πρέπει να σας διορθώσω, λέει ο πρόεδρος. Δεν θα είναι δύο οι αντιπρόσωποι. Ο αντιπρόεδρος ε, ακύρωσε και εκείνος ε, το ταξίδι του, πρόσωπο του Μάρτιν Σούλτς, ε, ούτε η αν δεν θα πάει, οπότε δεν θα πάει κανείς. Ε, Επιτροπή των Περιφερειών θα πάνε τρεις. Ε, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα πάνε σε ένα ξενοδοχείο, δεν ξέρω σε ποιο ξενοδοχείο σε, ή δεν ξέρω καν αν είναι ξενοδοχείο. Δεν είναι καν κανονικό ξενοδοχείο, από ό,τι κατάλαβα, σε καμιά πανσιόν θα είναι. Οπότε... Για αυτά τα οποία είπαν η Judith Μέρκη, ο Βιτόριο Πρόντι και η λυπή αυτό θα... τι θα κάνουμε, ή όλοι ή ένας μόνο. Ή, κανένα. ή κανένας. Αυτά αποκρισταλώνονται. Λοιπόν, τώρα στον κατάλογο είναι Μπελιέ και μετά ο Ριχαρτ Ζέμπερ και τέλος ο Καλ Χάιντ Φλόρεντ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τις περισσότερες παρατηρήσει που ακούστηκαν, κυρίω για το κόστος. Και υποστήριζω και εγώ αυτό το επιχείρημα να μην το παρακάνουμε με το κόστος. Υπάρχει το θέμα της αντιπροσωπευτικότητας. Κατάρχα για το ψήφισμα. Ήμασταν πολλοί οι συγητές του ψηφίσματος. Και η θέση του Κοινοβουλίου για το Ρίο Συνένα. Αρχικά ήμασταν πολύ υποψήφοι τον Απρίλιο του 2011, πριν από ένα χρόνο και πολλοί εισηγητές εξ ονόματος της μου υπέβαλαν α, τροπολογίες. Με, την, α, με το όραμα των οικολόγων. Φυσικά κάποιοι συμφωνούν με, με μας, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο από άλλους. Και θέλουμε σε αυτή τη σύνοδο κορυφής αυτές τις απόψεις να τις περάσουμε για την νομιμότητα του εισηγητή υπάρχει ένα πρόβλημα. Το είπε και ο κύριο Πρόντι. Δεν ξέρω κατά πόσο μα εκπροσωπεί όλου. Δηλαδή η δύναμη του Κοινοβουλίου και είναι η μορφία του. Και θα κερδίσουμε, θα κερδίσουμε αν είμαστε πραγματικά αντιπροσωπευτικοί. Θα έχουμε μεγαλύτερο ειδικό βάρο. Και για να το ξαναπώ, Δύσκολο μου φαίνεται να είναι απόν το Κοινοβούλιο στην συνδοκορυφή για να υποβάλει, για να μιλήσει για το ψήφισμα, το δικό του ψήφισμα. Με βάση τις τελευταίες επαφές που είχα με τη Βραζιλία και με άλλα κράτη, μπήκε επιτάπητο σε αυτό το ψήφισμα. Η θέση του Κοινοβουλίου, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ήταν η πιο φιλόδοξη θέση από όλες τις θέσεις που υποβλήθηκαν. Θέλω να πάμε εκεί πέρα με φωνή βροντερή και με πολλά άτομα για να έχουμε μεγάλο ειδικό βάρος. Ε, το είπατε, από την Κομισιόν θα πάνε 4-5 επίτροποι. Ε, εδώ και ένα χρόνο ψηφίσαμε το... Περάσ... Υποβάλαμε μάλλον το ψηφίσμά μας, το ψηφίσαμε τον Νοέμβριο. Ε, πώς γίνεται ένα μήνα πριν τη συνδοκορυφής που γίνεται μία φορά τα 10 χρόνια δεν έχει ακόμα κάνει τίποτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κάνει κρατήσεις και για να αποφασίσει τι θα κάνει με τη συνοκορυφή. Το λέω και στην Επίτροπο. Πώς γίνεται, πώς οργανωνόμαστε, πώς εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο, στη Συνδοκορυφή του Ρίου. Μπορούμε χάρη στο, στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο να βρούμε τα μέσα να μην επιβαρύνουμε πάρα πολύ το προπολογισμό του Κοινοβουλίου κρατώντας την αντιπροσωπευτικότητά μας, να μείνει ψηλά η αντιπροσωπευτικότητά μας και παράλληλα μην ξεχνάμε το ψήφισμα το προσυπέγραψαν πάρα πολύ. Καταλαβαίνω την ε, οργή σας. Το θέμα αυτό ε, απασχολεί και την Κομισιόν και η Κομισιόν έχει αντίστοιχα προβλήματα δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να προβλέψουμε, αλλάξανε άρδιν οι συνθήκες. Και πράγματι πρέπει να ρωτήσουμε τους οργανωτές αν ο σκοπός τους ήταν να έχουν καλεσμένους στη Βραζιλία ή όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μας έχει εξοργήσει όλους και εμένα προσωπικά. Αλλά οι τιμές είναι αυτές οι οποίες σε είναι γνωστές. Επί 10 και 600 ευρώ σε, σε ξενοδοχεία να πληρώνουμε το βράδυ για δωμάτια τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε καν, αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια διαμαρτυρία η οποία θα είναι ουσιαστική για τα θέματα αυτά. Ο κύριος Ζέμπερ. Κύριε Πρόεδρε, τρεις με τεσσερισήμιση εδώ πέρα η μερίσια διάταξη γράφει συζήτηση με την ε, Επίτροπο Κόνι Χέντεγκαρτ, η οποία βρίσκεται εδώ πέρα. Εγώ δεν ξέρω να αλλάξαμε την ημερήσια διάταξη, παρακαλώ να τηρηθεί. Είναι και αγενές προ την κυρία Επίτροπο. Τώρα να καθόμαστε να συζητάμε αυτά τα πράγματα, αυτό είναι η πρώτη μου παράκληση. Τώρα, αφού θέλετε να γίνει αυτή η συζήτηση, σωστά συμπεριφερθήκατε, το συζητήσαμε πολλή ώρα στου ε, συντονιστέ, εμένω στην απόφαση των συντονιστών, με αυτέ τι συνθήκες πρέπει να στείλουμε σαφές μήνυμα. Όποιος δεν το καταλαβαίνει πρέπει να αναρωτηθεί το τι θα γίνει. Σκεφτείτε, μία φωτογραφία ενός συναδέλφου στο Κόμπα Καμπάνα και δεν μας ξεπλένει ούτε... Δεν έχουμε συνεδρίαση, σκεφτείτε. Πώς θα πάτε, πάτε σε ψηφοφόρο και θα πείτε πλήρωσα 600 ευρώ για νύχτε που δεν έμεινα χωρί αίθουσα συνεδρίαση, χωρίς να κάνω τίποτα. Καλή τύχη σας εύχομαι. Επίση, είχαμε πει να πάει ο κύριο Χερμπραντή, ο οποίος είναι ο εισηγητής. Τώρα ακούω πω συνυπέγραψαν κι άλλοι και να πάνε όσοι συνυπέγραψαν, Μπελιέ, Φλόρεντ κτλ. Ε, πρέπει να αλλάξουμε νομίζω την απόφαση. Είτε και οι συνυπογράφοντε πέντε άτομα, ή ακολουθούμε το σύστημα Deont και στέλνουμε τον Carl Heinz Florence. Εδώ είμαι ανοιχτό. Αλλά αυτό είναι ο μέγιστο αριθμό που μπορούμε να δικαιολογήσουμε. Σα το λέω ανοιχτά. Αλλιώ δεν υπάρχει καμία απόφαση στην οποία θα συμφωνήσω. Σα συμφωνώ. Σωστά αποφασίσαμε, το εξηγήσαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Είμαστε και εκπρόσωποι του λαού, πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας. Σας ευχαριστώ ή αν υποδηματά το Προεδρείο δηλαδή έβγαλε τα συμπεράσματά του, δεν θα εκπροσωπηθεί. Θα ε, πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε και με την ε, κυρία Επίτροπο το παγκόσμιο κλίμα είναι σήμερα το, το θέμα μας ε, και οπωσδήποτε πρέπει να ασχοληθούμε και σε αυτό. Λοιπόν, τελευταίος λοιπόν ο Καλ Χάιντς Κοιτάξτε, ε, όταν μιλάμε τώρα αγένεια, δεν είναι αγένεια, είναι προβλήματα, πρέπει να τα συζητήσουμε. Εγώ χαίρομαι για το ότι είναι εδώ πέρα η κυρία Επίτροπος, έτσι, για να το μάθει ότι δεν μπορούμε να καταπιούμε τα, τα πάντα. Δεν θα ήταν και εγώ να ήμουν ε, εδώ πέρα το πρωί συντονιστέ, δεν θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Ε, αντί για ένας ίσως να ήταν κανένας Αλλά ποια είναι η ουσία για μένα. εδώ και τρία χρόνια στο Κοινοβούλιο υπάρχει ένα κίνημα κατά αυτών των αντιπροσωπιών. Το είδαμε στο Ντέρμπαν, το είδαμε στο Κανκούν, ε, το είδαμε σε άλλες χώρες, στην Κοπενχάγη, ε, υπήρχε πάντα μια αρνητική πτυχή και ε, σε αυτό πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν έχουμε σύστημα σε αυτά τα συστήματα. Το κάνουμε και στις αντιπροσωπείες ε, με τη ΣΥΠΑ. Φεύγουν, οι, κόβουν τους διερμηνείς, κόβουν τους βοηθούς, κόβουν τους ε, πάντες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι εντάξει, μπορούμε να πάμε με 600 ευρώ ή δολάρια, αλλά δεν αντιδράσαμε. Έπρεπε να έχουμε αντιδράσει πολύ νωρίτερα και ζητάμε την προστασία της Κομισιόν. Πρέπει να μεγαλώσουμε επιτέλους και να θέμε να κερδίσουμε επιτέλους αυτά τα ζητήματα. Γιατί, κοιτάξτε, οι άνθρωποι που δεν θέλουν να γίνουν αυτά τα ταξίδια δεν θα κερδίσουν. Πριν από 20 χρόνια όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση γελάγανε μαζί μας. Τα πετούσε στην ανακύκλωση η Κομισιόν τώρα έχουμε αρμοδιότητες, πρέπει να πηγαίνουμε σε αυτές τι παγκόσμιες διασκέψεις γιατί έχει συνέπειε αυτό το πράγμα που θα τις νιώσουμε και θα πρέπει να τα εξηγήσουμε αυτά τα πράγματα στην περιφέρειά μας. Εμείς εκλεγόμαστε, όχι η Κομισιόν. Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των βουλευτών. Πολύ μικρότεροι, βλέπετε, μικρότερες αντιπροσωπείε, χωρίς βοηθούς, χωρίς διερμηνείς, χωρίς προσωπικό και... Εντάξει, αγαπητέ Ρίχαρντ, εγώ είμαι σε κάθε διάσκεψη. Εάν είναι να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά, μπορούμε να πάμε κάπου και να πιούμε και μια μπυρίτσα ήσυχη. Δεν ανάγκη να παραδεινόμαστε λοιπόν στα πάντα. Πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας για να μην βασιζόμαστε σε τρίτους αλλά μόνο στον εαυτό μας να μην πω δε το τι θα έκανα εγώ στο ταξιδιωτικό μας γραφείο που θα είναι μπουρλότο κανονικά. Μόνο μία παρατήρηση. Δεν θέλω να αναφερθώ στα ορίο και τα προβλήματα του ορίο. Αλλά θέλω να υποστηρίξω αυτό που λέει ο Καρλ Χάιντς Φλόρενς. Ότι το κλίμα στο κοινοβούλιο είναι πάντα να διαβρώνονται συνέχεια τα δικαιώματα των βουλευτών και ότι τουλάχιστον συνδέεται με οικονομικά δικαιώματα περιορίζονται συνέχεια. Σας παρακαλώ λοιπόν όλους αυτούς που είναι εδώ παρόντες να απευθυνθείτε στην ομάδα σας και να δείτε πώς λειτουργεί η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τι καινούρια ξεφουρνίζει κάθε χρόνο η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Και γιατί καταφέρνει αυτή η Επιτροπή να αποσπά την πλειοψηφία. Πρέπει όλες οι πολιτικές ομάδες να συνειδητοποιηθούν για το θέμα αυτό. Γιατί αλλιώς πάμε για τα μπάζα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταλήξει να μην έχει ουσιαστικά κανένα προϋπολογισμό να κάνει τίποτα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εγώ δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής. Αλλά βλέπουμε κάθε μέρα ποιες είναι οι συνέπειες από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Κρήτον. είμαι σύντομος. Έχω πάει τρεις φορές ε, σε τέτοιες αντιπροσωπείες, δύο φορές πλήρωσα από την τσέπη μου. Και μία φορά ήμουν στην επίσημη αντιπροσωπεία Είναι σημαντικό να είναι παρόν το Κοινοβούλιο, να συνεισφέρει. Δεν είναι διακοπές, έχει ρόλο που πρέπει να παίξει σε αυτή τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, ε, αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει αντιπροσωπεία αυτή τη φορά ή αν θα στείλουμε πέντε ανθρώπους απλώς. Πάντως αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο. Εμείς θα πρέπει να στέλνουμε αντιπροσωπείες, να οργανωνόμαστε εν ευθέτω χρόνο όταν εισιτήρια και δωμάτια είναι φθηνότερα και θα πρέπει να έχουμε τον χαμηλότερο δυνατό, να ξοδέψουμε τα λιγότερα δυνατά λεφτά. Αλλιώς δεν θα συνδεθούμε καθόλου με τα δρόμενα και νομίζω ότι συνολικά θα χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, λέει ο Νομίζω ότι έχουμε συζητήσει αρκετά για την κατάσταση αυτή. Έχω λάβει υπόψη μου αυτά τα οποία λέει ο κύριος Φλόρενς, ότι υπάρχει και συστημικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Και εγώ μπορώ να σας πω μονάχα ότι θα ξεκινήσω μια ε, πρωτοβουλία με, την, ε, με, τους πρόεδρους των, ε, των κοινοβουλευτικών ομάδων, έχουμε με την ε, συνδίκη Λισαβόνα αποκτήσει πολύ περισσότερες αρμοδιότητες. Έχουμε αρμοδιότητα για διεθνείς συμφωνίες, είμαστε συνομοθετική επιτροπή σε πάρα πολλά θέματα και αυτά έχουν συστημικές συνέπειες. Οι συντονιστές έχουν πάρει μια απόφαση η οποία δεν μπορεί τώρα να έρθει. Η απόφαση ελήφθη, αλλά όλες οι επικρίσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί έχουν καταγραφεί από μένα και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί, σας το λέω. Έχω προτείνει διάφορες ε, ε, προτάσεις για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, τις ανέφερα στους ε, συντονιστές, αλλά η πλειοψηφία των συντονιστών είπε να στείλουμε ένα μοναχά άτομο και αυτό θα είναι ο, ο εισηγητής μας. Αλλά από συστημική άποψη εγώ σας υπόσχομαι ότι θα πάρω την πρωτοβουλία το θέμα αυτό να συζητηθεί και να μπει σε κάποια τροχιά ώστε τα πράγματα να γίνονται με τακτικό τρόπο και όχι να μας καταλαμβάνουν εξαπίνης κάθε φορά τα γεγονότα και να βασιζόμαστε και στην καλή θέληση, αν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, των ε, οικοδεσποτών μας ή αν θα πρέπει να ζητούμε βοήθεια από την Κομισιόν, σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποδεχτούμε να υπάρχει μια τέτοια έκρηξη των, ε, ε, του κόστους διαμόνης εκεί. Εν πάση περιπτώσει κλείνω το σημείο αυτό και καλωσορίζω την κυρία Κόνη Χέντεγκαρτ από την Κομισιόν. Πιστεύω ότι ήταν σημαντικό να συζητήσουμε τα θέματα αυτά για την τμήμα της εργασίας μας και αυτά, αλλά Παρακαλώ. Μήπως να... Ο κύριος Φλόρινς χωρίς... χωρίς μικρόφωνο. Να σε βοηθήσω μονάχα. Δεν είναι σαφές αν θα πάει ένας ή κανένας. Αυτό θα ήθελα να ξέρω. Εγώ είχα ζητήσει να μην πάει κανένας. Δεν ξέρω ποια είναι η απόφαση η οποία τελικά θα υποστηριχθεί. Εγώ μπορώ μονάχα, λέει ο πρόεδρο, να υποστηρίξω αυτό που αποφασίσαν σήμερα το πρωί οι συντονιστέ Οι συντονιστέ είπαν με πλειοψηφία ότι ένας μονάχα θα πάει από την Επιτροπή μας. Και αυτό σας το αναφέρω ως απόφαση των ε, συντονιστών. Αυτή είναι και η επιστολή η οποία πήγε στους αρμόδιους για τα θέματα αυτά, γιατί έπρεπε να στείλω την επιστολή αυτή και στο Προεδρείο. Λοιπόν, το μόνο που σας επαναλαμβάνω είναι αυτό το οποίο είπαν οι συντονιστές. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Και δεν μπορώ εγώ με δική μου πρωτοβουλία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ανατρέψω αυτήν την απόφαση. Και έρχομαι τώρα στο σημείο 23 της ημέρας διάταξης. Γιολάινεν, ξέρετε πολύ καλά, ως πρώην πρόεδρος της Επιτροπής μας, Ναι, χωρίς μικρόφωνο. Η Λίνα Μακέβαν. Θα πρότεινα μονάχα, κύριε Πρόεδρε, το εξή. Σήμερα το πρωί, μόλις είχαμε μάθει τα νέα, δεν είχαμε χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Νομίζω πρέπει να ακούσουμε την, την ε, κυρία Επίτροπο, αλλά εμείς έχουμε ακούσει την άποψη των συναδέλφων θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους και θα δούμε ποιες πολιτικές ομάδες θέλουν να πάνε ή να μην πάει κάποιο. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να συνεργαστούμε με τι πολιτικέ μα ομάδε για να σα πληροφορήσουμε μέχρι τι 5 η ώρα το απόγευμα. Ναι, μπορείτε να, να κάνετε μια σφιγμομέτρηση όσο θέλετε των βουλευτών. Αλλά εγώ έχω ακούσει την απόφαση των συντονιστών και μετέφερα την καταπλειοψηφία απόφαση των συντονιστών στα αρμόδια όργανα. αλλά αυτό σημαίνει τα πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να πληροφορήσουμε και το Προεδρείο. Τώρα, αν θέλετε με τις 5 η ώρα, μπορείτε να συζητήσετε με τα μέλη των πολιτικών σας ομάδων. Αλλά εμείς είχαμε ήδη την απόφαση των συντονιστών και γι' αυτό εγώ προτείνω να συνεχίσουμε με την ημέρησια διάταξή μας, γιατί έχουμε ακόμα μονάχα ε, περίπου μια ώρα με την κυρία Επίτροπο και τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε μαζί της είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικές αλλαγές που θα μας μεταφέρει εδώ η κυρία Επίτροπος. Για τρίτη φορά λοιπόν καλώς ήλθατε κυρία Χέντεγκάρτ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έχουμε πάρα πολλές ε, πρωτοβουλίες που αντιμετωπίσαμε αυτή τη χρονική περίοδο το, την έκθεση Chris Davis, το νοδικό χάρτη για οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακα, Έχουμε μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εμπορία εκπομπών. Έχουμε το πακέτο αυτό που αφορά το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Και όπως ελέγχθη, 30 δολάρια το 30 ευρώ ο τόνος του διοξιδίου του άνθρακος είναι η κρίσιμη τιμή. Και οι τιμές κινούνται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, 6 με 8 ευρώ τον ε, τόνο. Και υπήρξε και η πρόσφατη σύνοδος των Υπουργών Περιβάλλοντος και σας δίνω το λόγο και χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Καλώς ήλθες, Κόνι Χέντεγκάρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το θέμα που μόλις συζητήσατε, να σας δώσω μια ενημέρωση που μπορεί να σας ε, βοηθήσει να αποφασίσετε. Είπατε πολύ ότι η Κομισιόν στέλνει πέντε. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα με εσά. Και εγώ μείωσα τις αριθ... τον αριθμό της ημερών της παραμονής μου, ε, τρεις νύχτες μόνο. Ε... και η αντιπροσωπεία στη, στη Βραζιλία και η αντιπροσωπεία στην Υόρκη το έχουν Τη τις νέες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το έχουν θέσει αυτό το θέμα. Θα προσπαθήσω να, να είμαι σύντομη για να μην είναι μονόλογος. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το που, είμαστε, το που έχουμε φτάσει στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, η Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα κατάφερε να αποφασίσει τι θα κάνουμε την επόμενη περίοδο με βάση τις αποφάσεις που πήραμε στον Τέρμπαν. Ίσως ξέρετε ότι είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις. Ανακουφίστηκα τέλο πάντων την περασμένη εβδομάδα που αποφασίστηκε με απαρτία τι θα κάνουμε και 27 τι θα γίνει και με το 30%, η προσφορά του 30% είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα που στέλνουμε στους διεθνούς μας εταίρους. Ε, σε διεθνές επίπεδο πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά προφανώς. Ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να πάρουμε θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι ήσασταν στον Τέρμπαν, ξέρετε ότι για την επόμενη διάσκεψη του κλίματος να λύσουμε το θέμα με τον αέρα η επόμενη προεδρία είναι του Κατάρ. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα σχέδιο εργασία λειτουργικό, ούτω ώστε μέχρι το 2015 να έχουμε τη Διεθνή Συμφωνία. Δηλαδή, υπολογίζουμε ποιο θα πρέπει να έχει κάνει τι μέχρι το 2015. Ποια θέματα θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί, ούτω ώστε να μπορούμε εμεί να ολοκληρώσουμε τι διαπραγματεύσει για το νέο διεθνέ καθεστώ μέχρι το 2015. Παράλληλα. Υπάρχει και ένα κενό φιλοδοξία εδώ. 7 και 8 Μαΐου έχουμε προσκαλέψει φίλους από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για να κάνουμε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και για τον Τέρμπαν και για το τι θα γίνει μετά, ε, νόψη της Ντόχα, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί και για το Ρίο συν 20. Γιατί η συμμαχία που δημιουργήσαμε στο Δέρμπαν και πριν θα ήταν καλό να λειτουργήσει και εν ώψη του Ρίο τον Ιούνιο. Εκεί είμαστε λοιπόν, εκεί έχουμε φτάσει στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και αν σας ενδιαφέρει κάντε μου σχετικές ερωτήσεις. Τώρα, για τα εσωτερικά μας. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην άτυπη συνάντηση των ε, Υπουργών Περιβάλλοντος για πρώτη φορά στο Συμβούλιο συζητήσαμε το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ήταν πολύ ενθαρρυντικό το ότι όλα τα κράτη-μέλη, όλα, το τονίζω, αναγνώρισε ότι το σύστημα, αναγνώρισε το σύστημα αυτό ήταν και είναι και θα πρέπει να είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα. Ομόφωνα το αναγνώρισαν αυτό και είναι θετικό. Επίσης, ξεκάθαρο ήταν ότι πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα βραχυπρόθεσμα και κάποια πράγματα μακροπρόθεσμα. Ε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε από πλευράς κομισιών. Παράδειγμα χάρη, του, την αναθεώρηση του συστήματος ε, εμπορία εκπομπών ε, που θα την παρουσιάσουμε. Λέγαμε την παρουσιάσουμε το 2013, αλλά τελικά θα την παρουσιάσουμε ε, μέσα στο 2012 σε λίγους μήνες. Μέσω αυτής της αναθεώρησης μπορούμε να δούμε τι εναλλακτικέ λύσεις έχουμε σε ό,τι αφορά τις δημοπρατήσεις δικαιωμάτων. Πολλά δικαιώματα θα πρέπει να μπουν στην αγορά ε, για την περίοδο 2013 με 2020. Ενώ λίγες, λίγα δικαιώματα θα μπουν τα τελευταία χρόνια. Ε, και πώς αυτό θα επηρεάσει τις αγορές. Εκεί θα παρουσιάσουμε κάτι ούτως ώστε να έχουμε μια πρόταση για να ληφθεί απόφαση πριν από το τέλος του 2012. Αυτό είναι μια βραχυπρόθεσμη ιστορία. Αν θες να κάνεις κάτι με χαμηλές τιμές ETS, ε καλό είναι να θέσεις υψηλότερο στόχο. Δηλαδή να έχεις υπόψη σου ε, τι θα γίνει και μετά το 2020. Και από τις ε, ανεπίσημες ε, συζητήσεις με τους υπουργούς προκύπτει ότι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να έχεις και το μετά το 2020 υπόψη, χωρίς να παίζει με την αγορά. Έπειτα η διαπραγματεύση για την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Τι θα γίνει με το set aside. Και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για το μήνυμα που έστειλε και σας ευχαριστώ για την ε, ψηφοφορία στις 15 Μαρτίου για τον οδικό χάρτη για χαμηλές εκπομπές. Και ξέρω πολύ καλά ότι κυρίως η Επιτροπή σας δούλεψε πολύ για να το πετύχετε αυτό. Και στείλατε ένα διαπαραταξιακό ισχυρό μήνυμα, το οποίο λάβαμε. Τώρα, για να μην πολυλογώ. Άλλο θέμα. Αεροπλοεία. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Πάλι μιλάω για την ε, ψηφοφορία που έγινε μέσα Μαρτίου. Γίνονται πολλές συζητήσεις με πολλές χώρες που δεν τους αρέσουν η, νομοθεσία μας. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια ήδη τώρα για να δούμε πώς μπορούμε ε, να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα. Μετά από τη συνάντηση στη Ρωσία, ε, πολλές χώρες έχουν πιστεί ότι είναι καλύτερο το παγκόσμιο σύστημα. Είπαμε εντάξει, αλλά για να δούμε, μπορούμε να πετύχουμε ε, παγκόσμια συμφωνία μέσω της Διεθνού οργάνωσης. Ε, τον περασμένο μήνα αποφασίστηκε ότι οι μηχανισμοί αγοράς θα πρέπει να αναλυθούν εκ του σύνεγκης, Θα πρέπει να συζητηθούν στο Συμβούλιο ΙΚΑΟ τον Ιούνιο και ελπίζω μέχρι το φθινόπωρο να έχουμε μία ιδέα για το αν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει παγκόσμια συμφωνία. Υπάρχει βούληση ή δεν υπάρχει βούληση. Έχω δύο άτομα μόνιμοι, μόνιμους από την δική μου, το δικό μου γραφείο ε, και από την αρμόδια γενική διεύθυνση που προσπαθούν να πετύχουν να, να εξασφαλίσουν αυτή τη συμφωνία. Για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ξέρετε γιατί είναι σημαντικό για μας αυτό, ε, θα πρέπει τα κλιματικά θέματα να μπουν σε διάφορες γραμμές του προπολογισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην Κομισιόν πιστεύουμε ότι αν το πετύχουμε αυτό με την ενέργεια, ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, μεταφορές, αν δώσουμε πολύ πιο έξυπνα χρήματα στην κοινή γεωργική πολιτική, θα πετύχουμε ε, καλύτερα αποτελέσματα για τα λεφτά που ξοδεύουμε τους φορολογουμένων μας. Εσείς έχετε τα, τις απόψεις στο Κοινοβούλιο, αλλά μην ξεχνάτε ότι πολλές κυβερνήσεις προτιμούν την έννοια της ευελιξίας, που σημαίνει στείλε μας τα λεφτά και εμείς θα δούμε πώς θα τα ξοδέψουμε. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την ε, επαχθή οικονομική συγκυρία της Ευρώπης να αποδείξουμε ότι όταν στέλνουμε χρήματα εδώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα χρήματα δεν είναι σπατάλη, το κάνουμε για να υπάρξει ανάπτυξη, θέση απασχόληση, δραστηριότητα που τη χρειαζόμαστε και φέτο και τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γίνουν κάποια πράγματα, γίνουν τέτοιου τύπου πράγματα μέσω του προπολογισμού μα. Στι αρχέ του 2012 υιοθετήσαμε μια πρόταση επίση για το LULUCF, δηλαδή για τη χρήση τη γη, την αλλαγή τη χρήση τη γη και την δασοκομεία. Ε, και για τις εκπομπές των ε, αερίων του θερμοκηπίου στον ε, γεωργικό τομέα και στο δασοκομικό τομέα. Θέλουμε μία μεθοδολογία καταρχήν και αργότερα να ανεβάσουμε τον πύχη των στόχων. Είναι τεχνικό το θέμα, αλλά είναι σημαντικό, γιατί είναι προϋπόθεση για να πετύχουμε η γεωργία και η δασοκομεία να συνεισφέρει, ούτω ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας για τις υπόλοιπες προτάσεις που θα παρουσιάσουμε πριν ε, το καλοκαιρινό διάλειμμα. Πρόταση για τα, την νομοθεσία αυτοκινήτων και τα 95 γραμμάρια μέχρι το 2020. Ελπίζω να το κάνουμε αυτό γρήγορα και μετά ετοιμάζουμε το στόχο μετά το 2020. Ε, επίσης, την αναθεώρηση ΕΦΚΑΖ, όπως λέτε και στο ψήφισμά σας, θα παρουσιάσω μια πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα καύσιμα και μετά το φθινόπωρο και ελπίζουμε να, να υπάρξει μια παγκόσμια απόφαση για την εξάλληψη κάποιων επιβλαβών καυσίμων. Για τις εκπομπές της ναυτιλίας μας συζήτησαν να προετοιμάσουμε κάποιον κανονισμό αν υπάρχει μια προοπτική παγκόσμια συμφωνίας και κάνουμε μια αξιολόγηση αντικτύπου την προπαρασκευαστική δηλαδή εργασία και τέλος προετοιμάζουμε μια στρατηγική προσαρμογή της Ένωσης. Ίσως είδατε πως δημοσιεύσαμε ήδη το Climate Adapt, μια ιστοσελίδα, ένα εργαλείο για να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, προσαρμογής. Σημαντικό αυτό για τις περιφέρειες και τις πόλεις. Αυτό για να σας πω κάποια από τα ζητήματα που προκύπτουν, αλλά βεβαίως η βασική συζήτηση είναι το τι θα γίνει με τις κλιματικές πολιτικές μετά το 2020 και αυτό υπό το φως ε, του ενεργειακού οδικού χάρτη μέχρι το 2050, το ακούς οδικούς χάρτες, αλλά και τι θα γίνει με την οδηγία ενεργειακής αποτελεσματικότητας, που βεβαίως ελπίζω να μην ε, ε, την ε, νερώσουμε και εξασθενήσουμε πάρα πολύ γιατί θα δημιουργηθούν έτσι δουλειέ στην Ευρώπη που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Κόνη για την ε, δήλωσή σας αυτή. Τώρα θα κάνουν ερωτήσεις πρώτα οι συντονιστές. Ρίχαρτ Ζέιμπερ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο, την κυρία Χέντεκαρτ για την εικόνα των δραστηριοτήτων της που μας ε, έδωσε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι επιτέλους έρχεται μια πρόταση για τους ε, χλωροφθοράνθρακες και μιλάμε για face down και όχι face out. Επίσης ε, υπάρχουν και νέες πρωτοβουλίες για τον λεγόμενο Τώρα, για τις διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις ε, θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι νέες ε, εξελίξεις από τους μεγάλους εταίρους μας, η και Κίνα. Υπάρχει καμία κίνηση. Αυτά τα οποία διαβάζουμε στα διεθνή μήμη φαίνεται πως ειδικά στις ΙΠΑ δεν υπάρχει τίποτα και ούτε κανένα θετικό βήμα ακούμε από την Κίνα όσον αφορά την συζήτηση που προκαλεί μεγάλη νευρικότητα στην ε, βιομηχανία ε, για τα δικαιώματα τα... και τα δικαιώματα τα οποία θα αποσυρθούν λόγω των χαμηλών τιμών. Ισχύει κάτι τέτοιο ή θα ε, συνεχίσει να ισχύει το σύστημα εμπορίας εκπομπών όπως έχει αποφασιστεί, δηλαδή χωρίς αλλαγές έως το 2020 και τέλος. Έχω την εντύπωση, κυρία Επίτροπε, πως ε, πολλά λόγια λέει η Κομισιόν ε, στην κλιματική πολιτική χωρίς να τα εννοεί. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι γίνεται εντός της Κομισιόν και ειδικά τι σκέφτεται ο Επίτροπος Βιομηχανίας ε, δεν ξέρω αν μπορεί να ασκήσει ταυτόχρονα και αν θέλει να ασκήσει κλιματική πολιτική. Ευχαριστώ. Λίντα Μακάβαν, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κυρία Επίτροπε. Σα ευχαριστώ για την υπομονή που δείξατε με την Επιτροπή μα σήμερα το απόγευμα. Είναι φανερό ότι έχετε την υποστήριξή μα για τα δύσκολα θέματα που έχουν να κάνουν με την αεροπορία και την εφαρμογή του ETS, του συστήματο εμπορία. Και χαίρομαι που και οι Υπουργοί σας δίνουν την υποστήριξή τους γιατί πολλές φορές γυρίζουν στις χώρες τους και πάβουν να σας υποστηρίζουν. Ό,τι αποφασίζεται στις Βρυξέλλες υποσκάπτεται σε εθνικό επίπεδο. Αλλά αυτό είναι το εργαλείο που έχουμε, το ETS, ε το σύστημα εμπορίας και επομένως πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να κάνουμε κάτι για το, τη διαδικασία set aside από το 2013 και μετά όταν αρχίσει ο πληστηριασμός ε, δικαιωμάτων εκπομπών. Είναι δύσκολα λοιπόν τα πράγματα πολλές φορές από πολιτική έποψη και ιδίως στον τομέα της αεροπορίας. Ξέρουμε ότι, <clears throat> ξέρετε ότι ξέρουμε ότι δεν έχετε απόλυτη υποστήριξη από το Συμβούλιο για μία σειρά από θέματα. Για, τις, για τους ασφαλτικούς ε, για τις ασφαλτικές άμμους και την ε, εξόριξη από τέτοια θέματα παραδείγματος χάρη δεν είχατε την υποστήριξη από το Συμβούλιο και είναι πολύ καλό που μας αναφέρετε για το τι θα γίνει μετά το 2020, γιατί όλη μας η νομοθεσία δεν ξεπερνάει το 2020, αλλά το 2020 είναι πολύ κοντά. Η κλιματική μας νομοθεσία ξεκίνησε από τέσσερα χρόνια. Μόλις αρχίσαμε να προχωρούμε με το σύστημα εμπορίας, άμα θέλουμε να σκεφτούμε τι γίνεται με τα αυτοκίνητα τα οποία θα είναι ακόμα στον δρόμο, πρέπει να σκεφτούμε και επιπλέον τι θα γίνει πέραν του 2020. Είναι πιο δύσκολο να εξασφαλίσουμε ότι οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν για στόχους μετά από το 2020. Αν δεν το κάνουμε όμως ποτέ δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσουμε σε αυτή την ομάδα και σε αυτή την Επιτροπή να πετύχουμε <clears throat> αυτούς τους στόχους και θέλουμε να ακούσουμε και τις δικές σας προτάσεις. Ευχαριστώ Λίντα. Δεν είναι μακριά το 2020 ο Chris Davis για τους φιλελεύθερους. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστώ που έχετε καλύψει με τα εισαγωγικά σα σχόλια τόσο ευρύ πεδίο. Τρία σημεία πρώτα απ' όλα. Είδατε τι ειδήσει από το Bloomberg σήμερα που κάνα μια μελέτη για το επενδυτικό κόστο τη επίτευξη μια μείωση 30% μέχρι το 2020 είπαν ότι είναι περίπου 7 με 9 ευρώ το άτομο. Δύο καφεδάκια. 1,5 στην Ελλάδα ίσως. Το χρόνο. Εντάξει, αυτά για τον καφέ, αλλά αυτό λέει το Bloomberg και το κόστος της επίτευξης αυτού του στόχου. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι ορισμένες χώρες, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και το Βέλγιο, θα πληρώσουν λιγότερο εάν πάνε για ένα στόχο που είναι πιο φιλόδοξο όπως το 30% από ότι για να πάνε σε 20% γιατί θα αυξηθεί το κόστος των ε, δικαιωμάτων εκπομπής και έτσι αυτό θα τους αποδώσει χρήματα. Δεύτερο, ένα ερώτημα μονάχα. Το θέμα της ε, ε, συγκράτησης και αποθήκευσης του άνθρακα, του CCS. Ένας διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ενέργειας είπε χθες ότι θα έχουμε αυξήσεις της 6 βαθμούς Κελσίου μέσα στον 21ο αιώνα αν δεν αλλάξουμε την πολιτική μας και η συγκράτηση και αποθήκευση άνθρακα θα είναι σημαντικό στοιχείο αυτής της πολιτικής. Μέχρι το 2020 θα πρέπει να έχουμε ε, ήδη 40 τέτοια κέντρα, 60 μάλλον τέτοια κέντρα για τη συγκράτηση του άνθρακα, του διοξιδίου του άνθρακος. Προβλεπόταν να υπάρχει μια μεγαλύτερη χρηματοδότηση, αλλά τώρα φαίνεται ότι μόνο 1,5 δισεκατομμύριο για τη συγκράτηση και την αποθηκεύση του άνθρακα προβλέπεται. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Αυτό είναι ένα κύριο συστατικό τη πολιτική μα και θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι για να προωθήσουμε τα θέματα αυτά. Για τα αυτοκίνητα τώρα και τι ε, απαγορεύσει που έχουν επιβληθεί, έχει μειωθεί κατά 20% από τη βιομηχανία η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος και έχει αυξηθεί η αποδοτικότητα στη χρήση των καυσίμων. Λυπάμαι από αυτά που ακούω ότι οι φιλοδοξίε τη νομοθεσία που προτείνονται δεν είναι τόσο ψηλέ όσο θα θέλαμε να είναι. Οι... μηχανικοί έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια, οι μηχανικοί κινητήρων κτλ. για να προωθήσουν τα πράγματα εδώ και κάνουν καταπληκτική δουλειά. Σε σχέση επίση με τι απαγορεύσει. Όταν εισήχθη αυτή η τελευταία νομοθετική ρύθμιση, για τα, για τα ε, ημιφορτηγά, τα ε, αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στα 180 γραμμάρια ο, ο στόχος ο οποίος προτείνεται. Επομένως, οι φιλοδοξίες της νομοθεσίας ε, ήταν χαμηλότερες από αυτό που θα έπρεπε να είναι, γιατί μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερο. Θα μπορούσατε να το ελέγξετε αυτό και να μου δώσετε μια απάντηση. Thank you Ευχαριστώ, Chris. Μας Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την υπομονή που δείξατε. Έχω τέσσερις σύντομες αλλά δύσκολες ερωτήσεις για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε για κάποια απόσυρση δικαιωμάτων και υπήρχε πλειοψηφία στην Επιτροπή μας και ακύρωση μετά των δικαιωμάτων αυτών. Τώρα όμως ε, σας ακούω και μιλάμε για αλλαγή της διαδικασίας δημοπράτησης. Αυτό είναι άλλο πράγμα γιατί αν αλλάζει απλά η διαδικασία δημοπράτησης δεν μιλάμε πλέον για ακύρωση. Μπορεί να ξαναφέρουμε, μπορεί να έρθει πιο νωρίς η αναθεώρηση, αλλά υπάρχει ζήτημα του ότι θα γίνει και πολλές αγορές λένε πως το να αλλάξει μόνο το χρονοδιάγραμμα διαπραγμάτευσης δεν δίνει το σωστό μήνυμα πως ε, το σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι η βάση των πολιτικών μας. Μπορείτε να μας τα εξηγήσετε λοιπόν. Δεύτερον, ε, εμπορία εκπομπών και αεροπορία. Έχουμε πληροφορίες από την Κίνα πως θα φορολογήσουν, λένε, κάποια, κάποιο κομμάτι της αεροπορίας. Πώς το κρίνεται αυτό σε ένα ισοδύναμο μέτρο που μπορεί να επηρεάσει τη συζήτηση με τους Κινέζους. Τρίτον, αυτοκίνητα. Ναι, μπορείτε να φέρετε πιο νωρίς μία πρόταση, αλλά βεβαίως το βασικό είναι η ετικέτα, να ξέρουν ο καταναλωτής τι αυτοκίνητο αγοράζει. Και όταν είχε ξεκινήσει πριν από δύο χρόνια ήταν σημαντικό αυτό, να ξέρουν οι καταναλωτές τι αμάξι αγοράζουν. Γιατί υπάρχει lobbying κατά του να ξέρουν ε, οι καταναλωτές. Τέταρτον, Ρίο είναι 20 σύντομα. Στο Τέρμπαν βεβαίως η μεγαλύτερη επιτυχία της Ένωσης ήταν η συμμαχία αυτή ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρικανικής Ένωσης και των λοιπών χωρών. Τι μπορούμε να κάνουμε ε, για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί αυτή η συμφωνία στο Ρίο. Ευχαριστούμε. Τελειώσαμε λοιπόν με τους συντονιστές και τώρα θα, ακούσε, ακούσουμε την κυρία Επιτροπή. Ευχαριστώ για τον Ρίχαρτ Τζέιμπερ για την σταδιακή κατάργηση, το phasing down. Αυτό το οποίο βλέπουμε από την ανάλυση μας είναι πως εάν καταργήσουμε πράγματα, τότε υπάρχει ρήτρα πως πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική διαθέσιμη. Άρα θα είναι έτσι αργότερη η πρόοδος. Οπότε, από το λεγόμενο face down. Οπότε, εξετάζουμε αυτή τη στρατηγική, τη μείωση και όχι την κατάργηση, γιατί έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως και δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάποια ε, εναλλακτική. Συνολικά λοιπόν θεωρούμε πως το καλύτερο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα είναι με τη μείωση παρά με την κατάργηση. Και αυτό εξετάζουμε. Πολλοί από εσά ε, ρωτήστε για την αεροπορία και τη νέα αυτή κινέζικη πρωτοβουλία. Την τρίτη που μας πέρασε νομίζω το Κινέζικο Υπουργείο έβαλε στη σελίδα του ένα νέο φόρο αεροπορίας ε, και θα πήγαιναν, λέει, τα έσοδα σε κάποιο είδους κλιματική δράση. Ρώτησαμε λοιπόν την αντιπροσωπεία μας στο Πεκίνο να δει τι γίνεται το εάν είναι ισοδύναμα μέτρα. Μπορεί να μην είναι, αλλά το εξετάζουμε γιατί ήταν ενδιαφέρον ε, τα έσοδα αυτά να πάνε με κάποιον τρόπο στα του κλίματος για τις ΙΠΑ αν υπάρχει κίνηση υπάρχει μια θέληση για διάλογο θα έλεγα και μια έθεση να μην ε, κλιμακωθεί η κατάσταση μέσω ανακοινώσεων. Θα ήθελα να δω τον γραμματέα, τον Υπουργό Μεταφορών, είχαμε κάτι επαφές. Υπάρχει ουσιαστικός διάλογος, αλλά ο διάλογος γίνεται στον ΙΚΑΟ. Δεν αρκεί να λένε ναι, θέμε παγκόσμια συμφωνία. Πώς αν τα μέρη λένε αυτό το οποίο λένε από το 1997, που τελικά δεν έγινε τίποτα, τότε δεν θα έχουμε συμφωνία στον ΙΚΑΟ. Οπότε, εξαρτάται από το εάν θέλουν α, κάποια νέα κίνηση. Και το εξετάζουμε αυτό. Υπάρχει μια συνέντευξη στο Rolling Stone που δημοσιεύτηκε χθες ή σήμερα του Προέδρου Ομπάμα που ανέφερε και σε, αναφέρθηκε και στο κλίμα και λέει πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Ε, συμφωνώ. Ας δούμε λοιπόν αν υπάρχει κάποια κινητικότητα γιατί αυτό το οποίο κάνουμε στην αεροπορία είναι ένας λογικός τρόπος πρόοδου. Αλλά βεβαίω αν έχουμε συμφωνία στον ΕΚΑΟ τι καλύτερο. Αλλά σας διαβεβαιώ πως αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών οι υπηρεσίες μας, ε, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, ε, τρέχουν και αυτοί για να εξηγήσουν σε άλλους το τι διακυβεύεται. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω πως υπάρχει μια κατανόηση. Πολλοί από εσά αναφέρατε την απόσυρση κάποιων δικαιωμάτων και αυτό το οποίο είπε η Λίντα Μακάβαν. Η απόσυρση <laughs> και η απόσυρση και η δημοπρασία είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γιατί κοιτάμε λοιπόν τώρα το τι γίνεται με τη δημοπρασία. Γιατί η μεθοδολογία του να περάσει αυτό είναι απλούστερη, να το πω έτσι. Από το να ανοίξουμε ξανά την οδηγία και να αλλάζουμε τα πάντα. Οπότε, η δημοπρασία στη δημοπρασία μπορούμε να παρουσιάσουμε κάτι στην Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής και εκεί πέρα δεν απαιτείται ομοφωνία. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο μπορεί να γίνει γρήγορα. Όλα τα άλλα θα χρειαστούν καιρό. Αυτό το οποίο προτείνουμε τώρα με το προφίλ της ε, δημοπρασίας αυτό δεν σημαίνει πως δεν εξετάζουμε άλλα πράγματα και τα έλεγα στον πρόεδρο εδώ πέρα για τις συζητήσεις που είχαμε την πέμπτη που μας πέρασε. Ε, ήταν όμως πολύ επικοδομητική αυτή η συζήτηση. Είναι σαφές σε πολλά κράτη-μέλη πως ε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά το 2020. Είναι σημαντικό αυτό. Μπείτε στη σελίδα της Δανέζικης Προεδρίας, γιατί εκεί πέρα μας παρουσίασαν τέσσερις διαφορετικές δηλώσεις με βίντεο τους διευθύνοντες συμβούλους της ΣΕΛ, της Euroelectric, της Alstom και το Γενικό Διευθυντή της Business Europe. Και όλοι είπανε στις δηλώσεις αυτές προς τους υπουργούς σας παρακαλούμε τώρα, κοιτάξτε το 2030. Για εμάς στη βιομηχανία το 2030 είναι αύριο. Εμείς κοιτάμε ήδη πέρα από το 2020 θέμε προβλεψιμότητα. Ε, εδώ πέρα λοιπόν Πρέπει να το δούμε αυτό. Και ξέρουμε με τον οδικό χάρτη χαμηλών εκπομπών και τα λοιπά πως υπάρχουν προκλήσεις. Αλλά νομίζω πως όλο και περισσότερα κράτη-μέλη συνειδητοποιούν γιατί και η βιομηχανία μας ζητάει να κοιτάξουμε παραπέρα. Και μετά η συζήτηση για τη σταδιακή απόσυρση θα επανέλθει. Ελπίζω όταν συζητήσουμε την ε, οδηγία ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Και βεβαίως εξακολουθεί να είναι η θέση της Κομισιόν πως υπάρχει σχέση μεταξύ του τι προκύπτει από εκεί και τη συζήτηση της αδιακής απόσυρσης. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση με τα κράτη-μέλη και στο πλαίσιο της οδηγίας, αλλά ελπίζω πως ε, θα υπάρξει μια τάση απολογισμού και να γίνει αυτή η συζήτηση και πολλά κράτη-μέλη προς τα εκεί πήγαιναν. Ρωτήσατε για το ποιο είναι το κλίμα το, στην Κομισιόν, στον κλάδο κτλ. Στην Κομισιόν είναι πολύ σαφές ότι οι κλιματικές πολιτικές, η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όλο αυτό το πακέτο θεωρείται ως ε, Πηγέ δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην, ε, στην Ευρώπη. Ε, είδατε την περασμένη εβδομάδα και τη σχετική ανακοίνωση. Αυτή είναι οι, τρει τρεις που θεωρείται ότι μέχρι το 2020 μπορούν να δημιουργήσουν πολλές υγείες, πολλές θέσεις απασχόλησης. Πράσινη οικονομία, υγεία, μόνο η πράσινη οικονομία μπορεί να δημιουργήσει 6 εκατομμύρια θέσει απασχόληση. Και εκεί βλέπουμε πόσε θα προέλθουν από τι ανανεώσιμε, από την ενεργειακή αποδοτικότητα κτλ. Υπάρχει συμφωνία στην Κομισιόν ότι θα πρέπει να παίξει κεντρικό ρόλο στην δημιουργία θέσεων απασχόληση και ανάπτυξη. Γι' αυτό θέλουμε να την περάσουμε παντού και στον προπολογισμό, αλλά και στον, στην πρόταση του προπολογισμού για την καινοτομία. Τώρα, ο κλάδος είναι πιο διαιρεμένος. Αλλά θεωρώ ότι και μερικές από τις οργανώσεις των βιομηχάνων το συζητάνε πάρα πολύ έντονα, γιατί βλέπουν ότι σε πολλούς τομείς στην Ευρώπη χάνουμε θέσεις απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, ένας τομέας που αντιστάθηκε πολύ καλά στην κρίση είναι, ήταν ακριβώς η πράσινη οικονομία, οι σχετικές αυτές θέσεις απασχόλησης. Ε, δεν, είναι κάτι λοιπόν το μελλοντικό αυτή η ιστορία της πράσινης οικονομίας. Το είδαμε το... ανάμεσα στο 2008 με 2010. Υπάρχει και σχετικό έντυπο υλικό από τους υπουργούς που το αποδεικνύουν. Λίντα. Συμφωνώ με αυτά που είπες. Δεν αρκεί να μιλάμε για αυτές τις πολιτικές, θα πρέπει να πάρουμε και αποφάσεις. Τις αποφάσεις που χρειαζόμαστε. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να πείσουμε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν το έχουν συζητήσει ακόμα το θέμα οι Υπουργοί. Πριν το συζητήσουν, θέλουμε να δούμε τι θέση έχουν τα κρατημέλη μέσω μιας μελέτης επιπτώσεων, μέσω μιας μελέτης αντικτύπου, ούτω ώστε να ετοιμάσουμε την πρόταση για τους Υπουργούς, για να καταλάβουν ότι το θέμα δεν είναι έτσι, ένα μικρό πράγμα, είναι κάτι που έχει πραγματική σημασία. Αυτή είναι η άποψη της Κομισιόν. Chris Davis. Είδα το Bloomberg και τα έσοδα από το, τη δημοπράτηση α, και το θέμα αυτό που είπες. Όταν συζήτησαν το θέμα αυτό οι υπουργοί, κατάλαβαν ότι το σύστημα είναι οικοδομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε ε, να συνδέονται αυτά τα έσοδα με τα δικαιώματα για εκπομπέ. Συνειδητοποιούν αυτό το πράγμα και προσπαθούμε να το, να το πούμε και στους Υπουργούς Οικονομικών για την δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Έχουμε τα διάφορα project. Πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη να δουν ποιε προτεραιότητε έχουν και πώς κατανέμονται ένα project. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν από κοινού την προσπάθεια. Είναι μία από τις τεχνολογίες, δεν είναι η μόνη από τις τεχνολογίες, αλλά είναι μία σημαντική τεχνολογία και καλό θα ήταν να προχωρήσει η Ευρώπη για τα αυτοκίνητα. Ε, για τα 180 γραμμάρια και τα 203 γραμμάρια. Θα το ξαναδούμε. Για, τους, για τις αυτοκινητοβιομηχανίες το 2020 είναι πολύ κοντά. Ε, γιατί αυτοί προγραμματίζουν πολύ πιο μακροπρόθεσμα. Ε, απλώς εμείς βάζουμε εμείς το κουτάκι των 95 γραμμαρίων και για να δούμε τι θα γίνει μετά το 2020 για πιο φιλόδοξα φιλόδοξου στόχους. Έχουμε λοιπόν μια διτή προσέγγιση μέχρι το 2020 και μετά. Ετικετοθεσία. Συμφωνώ μαζί σου. Μετά από δυόμιση χρόνια σε αυτή τη θέση, δεν καταλαβαίνω γιατί δημιουργεί τόσες πολεμικές αυτό το θέμα πρέπει να κάνουμε πρωτοβουλίες, να τι προωθήσουμε από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές να έχουν νόημα για του πολίτες. Να δουν τι επιλογές έχουν. Καλό θα ήταν. Δεν καταλαβαίνω γιατί δημιουργεί τόσες, τόσα προβλήματα η ετικετοθεσία. Για το ΟΑΣΙΣ και το LDC, τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Θα το συζητήσω αύριο με τους συναδέλφους μου. Έχουμε προσκαλέσει αυτές τις χώρες, ε, τις λιγότερο ανεπτυγμένες, 7 και 8 Μαΐου. Όταν τελειώσουμε τις συζητήσεις το βράδυ της 8 Μαΐου, ελπίζω να έχουμε ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα. Να πούμε, να τρία-τέσσερα θέματα, θέματα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάποιες άλλες χώρες και κάποιες λιγότερες ε, ανεπτυγμένες, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μπορούμε κάτι να βγάλουμε από το Ρίο. Ε, η ατζέντα του Ρίο είναι πολύ ευρεία. Τουλάχιστον να δούμε σε ποια σημεία μπορούμε να χτίσουμε συμμαχίες και αν τις χτίσουμε αυτές τις συμμαχίες κάτι θα αλλάξει για το Ρίο και κάτι θα πετύχουμε. Γι' αυτό λοιπόν τους προσκάλεσα σε αυτή τη συνάντηση 7 και 8 Μαΐου. Ευχαριστώ πολύ Κόνη. Μας, είπες, ε, είπαν στην αρχή ότι έπρεπε να φύγει στις 4 ε, και 4. Μπορούμε να έχουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων όμως. Λοιπόν, έχω τον Καλ Χάιντς Φλόρενς, τον Γιώ Λάινερ, τον Μαζένης, Μέρκης, τον Αρσένη, τον Μέρκης και, τα... και τον ε, Ρωμάνο Πρόντι. Ο, ο γιο. Γιατί πρέπει να, σύντομα παρακαλώ, πρέπει να φύγει η Επιτρόπος. Ναι, πιστεύω ότι έχουμε μια ε, νέα μορφή, μια ανανέωση για τα καύσιμα, ε, όπως βλέπουμε τα καύσιμα των πλοίων κτλ. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ταιριάζει με την κλιματική πολιτική, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά αυτή η διαδικασία του fracking στις ΗΠΑ, η εξόριξη φυσικού αερίου και πετρελαίου από σύστολτους πηγαίνει προς την άλλη κατεύθυνση. Για τον άνθρακα επίσης, είδα την έκθεση για το σύστημα εμπορίας τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεπεράσουμε το μπλοκάρισμα από τη μεριά της Πολωνίας είναι το επόμενο ερώτημα. Ο Κρήτον έχει το λόγο. Thank you very much. Uh, very briefly in Durban we said we... Για τον Durban είπαμε ότι θα ε, δεσμευτούμε αν μας δώσετε ένα οδικό χάρτη. Μας δώσανε αναπτυσσόμενες χώρες ένα οδικό χάρτα, χάρτη, αλλά αυτό ήταν μονάχα μια πολιτική δέσμευση χωρίς τροποποιήσεις για το πρωτόκολλο του Κιώτο. Είναι το έτος της αλήθειας τώρα τόσο για το Κιώτο και για τους ε, συμμάχους μας. Είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευτεί και να δεχτεί τροποποίηση στο πρωτόκολλο του Κιώτο, στο Κατάρ. Ποια είναι η στρατηγική μας, ποια είναι η δυναμική που διαγράφεται αυτή τη στιγμή και αν υπήρξαν κάποιες ε, διαμαρτυρίες από τους συμμαχούς μας για το γεγονός ότι δεν καταθέσαμε μια πρόταση που να περιέχει τροπολογίες. Κυρία Γκαρντίνη, συγγνώμη. Να επανέλθουμε στο σύστημα ETS, εμπορίας εκπομπών. Ε, κατάλαβα ότι κάτι θα κάνετε, αλλά δεν κατάλαβα τι θα κάνετε. Αν μία από τις υπόθεσεις είναι να παγώσουμε ποσοστώσεις, τι θα τις κάνουμε τελικά, πού θα καταλήξουν αυτές οι ποσοστώσεις. Αλλά κυρίως θέλω να μάθω τι, είναι, τι σκοπεύετε να κάνετε για να προστατεύσετε την ευρωπαϊκή βιομηχανία από τον κίνδυνο της διαρροής των εκπομπών. Μέρκες. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για όλα όσα μας είπατε. Δύο ερωτήσεις. Για τη διαφάνεια. Για τις ε, αιτήσει, ε, για ε, δωρεάν δικαιώματα εκπομπής, για τις εταιρείε παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Πολωνία, ένας υπάλληλος κομισιόν ζήτησε ε, στοιχεία για, θα, για αυτές τις αιτήσει. Εμείς δεν μπορέσαμε να τις δούμε. Πώς μπορούμε να δούμε αυτά τα στοιχεία και πότε μπορεί και το κοινό να ξαναδεί αυτά τα, τις αιτήσει για δωρεάν δικαιώματα εκπομπών. Ένα άλλο πολύ συγκεκριμένο ερώτημα αφορά την ουδετερότητα του άνθρακα των εκπομπών. της βιομάζας. Με βάση τους σημερινούς κανόνες δεν κάνουμε διάκριση ανάμεσα κατάλοιπα ξύλου και της βιώσιμης βιομάζας. Θεωρείται και τα δύο ουδέτερα. Θα το αλλάξετε, Κομισιόν, αυτό το στοιχείο. Ευχαριστώ, Ο Βιτόριο. Please, Vittorio, short. Ευχαριστώ, Επίτροπε. θεωρείτε ότι είναι πιθανόν οι ΙΠΑ να επικυρώσουν το πρωτόκολλο του Κιώτο. Είναι μάλλον απίθανο, θεωρώ εγώ. Και εν αυτή περιπτώσει υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν συμφωνίες ούτως ώστε από το δικό μας πρόγραμμα, να, μάλλον το δικό μας πρόγραμμα και το πρόγραμμα των Ηνωμένων κάπως να συγκεραστούν. Και δεύτερον, η απόφαση της Κίνας Πού εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, μπορεί να έρθει να κάνει το, τη μισή διαδρομή προς ε, ένα σύστημα ETS η Κίνα. Εικόνη. Συγγνώμη, πρέπει να είμαι πάρα πολύ συνοπτική τώρα για το αέριο από τις ασφαλτικές άμμου. Κοιτάμε τώρα, υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό. Εξετάζουμε το κατά πόσο η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επαρκής ή αν θα πρέπει να υπάρξουν ειδικοί κανονισμοί για τη διαδικασία της, ε, του κατακαιρματισμού του φράκινγκ για την εξόριξη αερίου. Επίσης, την υδρορογμάτωση. Για την Πολωνία. Πιστεύω ότι η Πολωνία ενδιαφέρεται να προχωρήσει για τα θέματα αυτά του, της χρήσης άνθρακα και τους ενδιαφέρει και η απόδοση ενέργειας. Οι όχι μόναχα εισάγουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία, αλλά εισάγουν και πάρα πολύ άνθρακα. Ξεχνάνε πολύ ότι συμβαίνει αυτό στην Πολωνία. Υπάρχει αυξανόμενη λοιπόν ε, συνειδητοποίηση για το ρόλο της ε, απόδοσης για την ενέργεια και γι' αυτό κάνουν κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουν μια μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην ενέργεια. Είχαμε λοιπόν μια πολύ σημαντική και πάρα πολύ επικοδομητική συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα και η Πολωνία υποστηρίζει πάρα πολύ και το σύστημα ε, εμπορία εκπομπών, το ETS. Ε, δεν πρέπει λοιπόν να, μην, να υπερβάλλουμε για τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για τον Κρήτονα, Αρσένη. Για το πρωτόκολλο του Κιώτο, ναι. Υπάρχει κάποια ισορροπία μεταξύ του να δώσουμε αυτά τα οποία είχαμε δεσμευτεί να κάνουμε στον Durban και στις, και στις δύο πλευρές. Δεν έχουν γίνει ακόμα όλα αυτά. Θα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη δεύτερη περίοδο δέσμευση στην Τόχα και όταν λες για άλλες ε, διαμαρτυρίες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, θα θέλανε να ε, επικυρώσουμε αμέσως τη δέσμευση αυτή, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στα άλλα πεδία. Αλλά πρέπει να πω επίσης ότι κατά τη δική μου άποψη αναγνωρίσουν απόλυτα και κατανοούν ότι πρέπει να εξευρεθεί μια ισορροπία μεταξύ αυτού που κάνουμε εμείς και του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε την πίεση για να κάνουν και οι άλλοι τα απαιτούμενα, χάρη σε σχέση με την ε, συμφωνία το 2015. Κυρία Γκαρντίνη, ίσως θα πρέπει να σας στείλουμε και ένα έγγραφο που αφορά τις διάφορες αυτές επιλογές. Ναι, είναι τεχνικά και είναι πολύπλοκα τα θέματα αυτά. Δεν θέλουμε να παγώσουμε τα δικαιώματα εκπομπή. Αλλά με τον τωρινό κανονισμό, αν δεν τον αλλάξουμε, θα υπάρχει τόσο υψηλό επίπεδο δικαιωμάτων που θα προκύπτει από το 2013 και 2014 και μόνο λίγα δικαιώματα θα περάσουν στην τελευταία περίοδο δημοπρασίας στη βιομηχανία. Και ρωτάμε αν είναι λογική αυτή η καμπύλη. Ίσως είναι καλύτερα να έχουμε λιγότερες, ε, λιγότερα δικαιώματα τα πρώτα χρόνια και μετά να προσθέσουμε όταν έχουμε ήδη αρκετά. Ο λόγος που τίθεται αυτό το θέμα είναι ότι οι εταιρείε μπορούν ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουν τις, ε, τα δικαιώματα αυτά σαν ένα στοιχείο εγγύησης στις τράπεζες. Μπορούν κατά κάποιο τρόπο να τις εκμεταλλευτούν. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο φυσιολογικό επίπεδο τιμών. Λόγω του συστήματος με τον οποίο μπορούν να εμπορευτούν τα δικαιώματα οι εταιρείε μπορούν να συνεχίσουν να είναι πολύ Χαμηλέ οι τιμέ των δικαιωμάτων εκπομπών ακόμα και όταν οι δραστηριότητε των βιομηχανιών έχουν επανέλθει σε φυσιολογικό επίπεδο. Με τέτοιε προκλήσει, λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε αν θα πρέπει να πλημμυρίσουμε την αγορά με με περισσότερα δικαιώματα που κινδυνεύουν να χαμηλώσουν ακόμα περισσότερο τις τιμές των δικαιωμάτων. Θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο οι διαφορετικές αλλαγές και πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό περισσότερο σε λεπτομέρεια και με τα κράτη-μέλη, αλλά αυτό ακόμα, ακόμα είμαστε στο επίπεδο ανάλυσης των διαφόρων επιλογών. Για την κυρία Μέρκης, για τη βιομάσα, έχουμε το κριτήριο βιωσιμότητας, το οποίο το αντιμετωπίζει η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του κυρίου Έττιγκερ, και έχουμε παρουσιάσει αυτή την πρόταση η Λουσιεφ, η οποία θα μας δείξει πώς μπορούμε να έχουμε ακόμα πιο βιώσιμη χρήση της βιομάζας για τα δωρεάν δικαιώματα στα κάτι μέλη. Είναι δική τους κρίση αν θέλουν να δημοσιοποιήσουν τι έχουν ζητήσει μορφή αιτήσεων από την Κομισιόν. Εμείς ενθαρρύνουμε τα κάτι μέλη να τα κάνουν όλα αυτά δημόσια και πολλά κάτι μέλη το έχουν κάνει, αλλά προτίμησαν να μην τα δημοσιοποιήσουν γιατί λένε ότι θα πρέπει να προστατεύσουν πληροφορίες που είναι ευαίσθητες για τις ενεργειακές τους εταιρείες. Η δική μα τάση πάντω ήταν να του ενθαρρύνουμε, αλλά δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να δημοσιοποιήσουν αυτέ τι πληροφορίες. Και κύριε Πρόντι, δεν κατάλαβα πολύ καλά το ερώτημά σα. για το αν οι Αμερικάνοι θα χειρώσουν το Κιώτο. Φυσικά μάλλον η απάντηση είναι όχι. Πρέπει όμω να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα μελλοντικό καθεστώ. Κάναμε τα πρώτα βήματα για αυτό στον Τέρμπαν. Συγγνώμη που ήμουν τόσο σύντομη, αλλά θα έπρεπε ήδη να είμαι κάπου αλλού θα ήταν πολύ άσχημο να αργήσω εκεί για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κλιματικά θέματα. Κόνη, σε ευχαριστούμε. Εντυπωσιάστηκα. Είσαι μαραθωνοδρόμος. Και νομίζω πως ε, έχεις ε, ανεξάντλητη ενέργεια, παλεύεις για την ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική και είσαι δραστήρια. Θα έχει τη στήριξή μας ε, την πλήρη στο μέλλον, στην νομοθετική διαδικασία Κασία, Το σύστημα μπορεί να κουμπώνει η βάση της κλιματικής μα πολιτική και μπορείς να συνεχίσει. So, jetzt geht's weiter. Και συνεχίζουμε. Με το σημείο 24. Εφαρμογή τη θεματικής στρατηγικής Η εφαρμογή θεματική στρατηγική για το έδαφο. Προτείνω να ακούσουμε πρώτα απ' όλα την Κομισιόν και μετά πάμε τη συζήτηση. Good afternoon, Mr. Chairman. My head of unit was supposed to be here, but I can, I can start on this point. Ευχαριστώ. Ο τμήματάρχης μου απουσιάζει. Ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την έκθεση για την εφαρμογή της θεματικής στρατηγικής για το έδαφος που ευθύθηκε πριν από πέντε χρόνια και θα θέλαμε να παρουσιάσουμε άρα μια ενημέρωση για την πρωτοβουλία αυτή και να καταδείξουμε την πρόοδο ή την έλλειψη αυτής για την προστασία του εδάφους ε, της Ένωσης. Μία έκθεση που συνοδεύεται μια τεχνική έκθεση από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Κομισιόν με λεπτομερείς πληροφορίες για την κατάσταση του εδάφους στην Ευρώπη στον βαθμό που έχουμε δεδομένα. Και η υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται στην Ευρώπη. Χάνουμε γη λόγω της αστικής ανάπτυξης των υποδομών, οι εκτιμήσεις μας και μιλάμε για συντηρητική εκτίμηση του προβλήματος είναι πως τουλάχιστον 270 εκτάρια γης χάνονται λόγω της ε, Ανάπτυξη των πόλεων και των υποδομών κάθε μέρα, δηλαδή μιλάμε για χίλια τετραγωνικά χιλιόμετρα το έτος. Κάθε 10 χρόνια δηλαδή ε, μία έκταση σαν την Κύπρο. Ή αν θέλετε μια άλλη σύγκριση, η συνολική επιφάνεια, μάλλον η συνολική καλλιεργήσιμη γη της Ολλανδίας, η συνολική αρωτρέα γη. Μιλάμε, αυτό το οποίο λέμε δηλαδή σφράγισμα του εδάφους από ένα διαπέραστο στρώμα εδάφους. Ε, επίσης έχουμε διάβρωση, 1,3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα που επηρεάζονται από τη διάβρωση. 20% αυτών ε, υπερβαίνει τις βιώσιμους ρυθμούς. Ε, υπάρχει πρόβλημα αλάτωσης του νερού λόγω των ε, τακτικών ε, άρδευσης. Ε, επίσης υπάρχουν προβλήματα ρήπανσης του εδάφους, αλλά βεβαίως δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αλλά υπολογίζουμε πως υπάρχουν γύρω στα 3 εκατομμύρια πιθανώς μολυσμένα σημεία στην Ένωση, 250.000 από τα οποία ε, θέτουν σοβαρό σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Οπότε όλα αυτά επηρεάζουν την δυνατότητα παραγωγής τροφίμων, αλλά έχει και υψηλό κόστος. Στην αξιολόγηση αντικτύπου η Κομισιόν υπολογίζει πως το συνολικό κόστος είναι γύρω στα 38 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο η διάβρωση κοστίζει 53 εκατομμύρια το έτος Οπότε δεν είναι μόνο θέμα του να αγαπάμε το περιβάλλον, έχουμε και κόστος ε, που επιβαρύνει την κοινωνία. Η κατάσταση, η ανάλυση που κάναμε το 2006 ε, δεν διαφέρει πάρα πολύ από αυτά τα οποία παρουσιάζουμε σήμερα. Η ανάλυση αυτή τότε οδήγησε στη στρατηγική αυτή που περιέχει μια πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο για το έδαφος και την προστασία του. Εγκρίθηκε μια πρώτη ανάγνωση λοιπόν από το Κοινοβούλιο το 2007. Τώρα είμαστε σε επαφή με το Συμβούλιο γιατί υπάρχει μια μειοψηφία που μπλοκάρει για να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν πως η στρατηγική αυτή είναι ένα συνολικό πακέτο. Υπάρχουν τέσσερις πυλώνες. Οι τρεις άλλοι είναι ενημέρωση, έρευνα το να ολοκληρωθεί σε άλλες πολιτικές. Ο τέταρτος πυλώνας είναι η νομοθεσία της Ένωσης ε, που είναι εξίσου ε, σημαντικός. Σύντομα, επίσης, να πω το εξής. Το τι έχει κάνει η Κομισιόν για να ενσωματώσει αυτά τα θέματα στις άλλες πολιτικές. Παραδείγματο χάρη, στην πρόταση μεταρρύθμισης κοινή γεωργικής πολιτικής ε, προτείνουμε σε πολλαπλές, ε, νέα πολλαπλή συμμόρφωση με την υποχρέωση να μην ε, οργώνουμε υγροτόπους και στη νέα πρόταση στηρίζουμε ρητό στην βελτιωμένη διαχείριση εδαφών για την δέσμευση άνθρακα και στη γεωργία και στην δασοκομεία. Τέλος, το πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα, όπως προτείνεται από την Κομισιόν της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπου ελπίζουμε να υιοθετήσει ο νομοθέτης, θα οδηγήσει σε βελτίωση της κατάστασης. Μια άλλη εξέλιξη των τελευταίων πέντε ετών ήταν η υιοθέτηση της οδηγίας βιομηχανικών εκπομπών μετά την οδηγία IPPC με διατάξεις για να διασφαλίσουμε πως η λειτουργία μιας βιομηχανικής εγκατάστασης δεν επιδεινώνει την ποιότητα του εδάφους. Προσπαθήσαμε λοιπόν να θέσουμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής για την νέα ρήπανση. Όμως υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις ε, που δεν καλύπτονται και βεβαίως υπάρχει και η κληρονομιά του παρελθόντος που δεν ε, υπόκειται στην οδηγία τρίτο στοιχείο όσον αφορά την ενσωμάτωση στις άλλες πολιτικές είναι χρηματοδότηση ειδικά για τα μολυσμένα σημεία και στην τωρινή περίοδο χρηματοδότησης 2007-2013 υπάρχουν γύρω στα 3 δις ευρώ διαθέσιμα για αυτή τη δουλειά και η διαπολιτική πολιτική θα συνεχιστεί για την αναζωογόνηση των σημείων αυτών. Τρία σημεία θέλω να τονίσω, ε, ιδιαίτερη σημασία που προκύπτουν από την έκθεση. Ένα, όπως ανέφερα, είναι η έλλειψη δεδομένων. Δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες ε, πάντα για να αξιολογήσουμε πλήρως την κατάσταση όσον αφορά την ε, εξέλιξη του εδάφους στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε σκεφτόμαστε έρευνες σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω τηλεπισκόπησης για να βελτιωθεί η γνώση που έχουμε δεύτερον. Όπως είπα, η ε, κάλυψη των εδαφών, όπως σας είπα κάθε 10 χρόνια χάνεται ε, έδαφος ε, ίσο με την έκθεση της Κύπρου και στον οδικό χάρτη η Κομισιόν είχε πει πως μέχρι το 2020 η πολιτική μας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο ρυθμός ε, αυτής της κατάστασης ε, θα πρέπει να έχει φτάσει μέχρι το 2050 να είναι μηδενικός. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε ένα μη δεσμευτικό ενδεικτικό κείμενο που περιέχει κατευθυντήριες γραμμές για την ε, αντιμετώπιση του σφραγίσματος του εδάφους και μειώνοντας ε, τον, τον αντίκτυπο του ανθρώπου. Κατόπιν υπάρχει και το όριο συνήκωση, μου απασχολεί αυτόν τον καιρό. Στην έκθεση πολιτικής ε, υπογραμμίζουμε πως η ανάπτυξη, η αύξηση του παγκοσμίου πληθυσμού και της κατανάλωσης ε, στις ανερχόμενες οικονομίες, η βιομάζα που χρησιμοποιείται για ενέργεια, όλα αυτά θα οδηγήσουν σε παγκόσμια χρήση της γης και πιθανή επιδείνωση της κατάστασης του εδάφους. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς λόγω πιθανών γεωπολιτικών ανισορροπιών αλλά επίσης γιατί θα εξαρτηθούμε ακόμη περισσότερο από τους σπόρους, τους εδαφικούς της Ένωσης, εάν ο κόσμος ε, φτάσει όπως αναμένεται τα 9 δισεκατομμύρια το 2050. Ε, Αυτός είναι ένας λόγος ε, για τον οποίο προτείναμε στην Σύνοδο Ρίο 20 το ζήτημα αυτό της υποβάθμισης του εδάφους θα πρέπει να είναι ένα από τα πέντε βασικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να επιτύχουμε αποτελέσματα και προτείναμε όλος ο κόσμος να συμφωνήσει με μηδενικό ρυθμό υποβάθμισης του εδάφους ε, σε κάποιο παγκόσμιο χρονικό πλαίσιο για να εστιάσουμε την προσοχή του κόσμου στις, πόρους τους εδαφικούς όχι μόνο όσον αφορά την ξηρά και τα πιο ξηρά εδάφη και αυτά που κινδυνεύουν με απερίμωση. Αλλά γενικά. Επίσης, σε δυο 3 εβδομάδες, 10-11 ε, Μαΐου, οργανώνουμε μία διάσκεψη για την αποκατάσταση και το σφράγισμα του εδάφους. Για κάποια από τα σημεία που ανέφερα δηλαδή. Είστε όλοι προσκεκλημένοι επί τη ευκαιρία η διάσκεψη θα κλείσει με μια συζήτηση με τον Επίτροπο Ποτότσνικ, Σιόλος, ε, εκπρόσωπο της Επιτροπής των Περιφερειών, το Γενικό Γραμματέα της Κοπακοτζέικα και ελπίζουμε εκπρόσωπο της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας. Έχω τρεις ομιλητές, ο Καρλ Χάινς Φλόρενς, η κυρία Χάουκ, και μετά ο Βιτόριο Πρόντι. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είχα αποφασίσει να είμαι ευρωβουλευτής και όχι να είμαι βουλευτής στο Βερολίνο στο, στην Bundestag γιατί τα θέματα της ε, υγείας και, της, ε, και του περιβάλλοντος ήταν τα θέματα που με ενδιαφέραν. Όλα αυτά τα οποία ακούω με κάνουνε να νιώθω κάποια ανησυχία. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουν να κάνουν με την ποιότητα του εδάφους τελικά έχουν αρνητικό αποτέλεσμα. Είναι αντιπαραγωγικά παρά το γεγονός ότι υπάρχουν οι κανόνες οι ευρωπαϊκοί. Είμαι γεωργός. Ξέρω ότι παραγωγός χάρη οι φυτογειονομικοί κανονισμοί περιέχουν κάποιες δοκιμασίες για το περιβάλλον που έχουν αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου. Αλλά όταν ζητάει κανείς να έχει μια πραγματική απάντηση για το τι γίνεται για την εφαρμογή αυτών των κανόνων, τίποτα δεν κάνετε για την προστασία των φυτών. Απολύτως τίποτα. Τι κάνετε για τις δοκιμασίες βιωσιμότητος στο περιβάλλον. Μα δεν έχετε ούτε καν καταλήξει σε ένα ορισμό του τι είναι κάτι που είναι βιώσιμο για το περιβάλλον εσείς κάνετε μια προσωμείωση για το τι γίνεται σε μια σειρά χρόνων. Μα είναι αυτό σωστό για τη βάση. Έχετε 15 κανονισμούς που ασχολούνται με τα θέματα του περιβάλλοντος. Το θέμα είναι όμως ότι κανένας από αυτούς δεν έχει πραγματικό αποτέλεσμα και δεν κάνουμε τίποτα για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που γίνονται στο περιβάλλον και αυτούς οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον. Εσείς λέτε ότι θέλετε μεγαλύτερο πλαίσιο για όλα αυτά, αλλά δεν μπορείτε να ελέγξετε ούτε μία οδηγία την οποία έχετε περάσει σε σχέση με, το, με τα εδάφη. Η οικογένειά μου δουλεύει τη γη εδώ και 30 χρόνια. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να φύγουμε από εκεί. Δεν θέλουμε ποτέ να μας πάρει την γη οι αρχές των Βρυξελών ή οποιοδήποτε άλλος. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό οι αρχές της Βόρειας Ιουνανίας Βεσφαλία και να λειτουργήσει η επικουρικότητα. Δεν πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να καταταγεί σε ομάδες κρατών ή πολιτών ή περιφερειών, οι καλοί, οι μέτροι και οι κακοί και να πείτε ότι αυτά τα εδάφη είναι καλά και εκείνα είναι λιγότερα, λιγότερα καλά. Και δεν μπορείτε να οργανώσετε ένα τέτοιο σύστημα για μεταφορά πόρων για το οποίο δεν θα υπάρξει ποτέ καμία α, πλειοψηφία. Πρέπει να βασιστούμε στην αρχή του ότι ο ρηπαίνων πληρώνει. Εμείς ε, ξέρουμε ότι έχουμε απογοητεύσει τον αρμόδιο επίτροπο για τα θέματα αυτά, γιατί εμείς αντιδρούμε σε αυτούς τους κανόνες που θέλετε να επιβάλλετε. Καταρχήν, θα πρέπει η στρατηγική την οποία έχετε ε, αναπτύξει να πετύχει ένα στόχο, γιατί αυτό το οποίο κάνετε δεν πετυχαίνει το στόχο του. Δεν έχετε επιτύχει τίποτα με ένα κανονισμό ο οποίος λειτουργεί ήδη για 10 και παραπάνω, 10-12 χρόνια. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απαγορευτεί και στην περιοχή που είναι το τριεθνές μεταξύ Γερμανίας, Ολλανδίας και Βελγίου βρίσκουμε στο νερό συνέχεια ουσίες οι οποίες είναι απαγορευμένες. Λοιπόν, βρείτε κάποιο τρόπο να ελέγχετε καλύτερα αν θέλετε να μιλήσετε για ποιότητα εδαφών. Και ήθελα να πω επίσης κάτι από την κυρία Βάισμπεργκερ, η οποία είναι η εμπειρογνώμη για τα θέματα αυτά και θα έλεγε και περισσότερα. Αλλά αυτά ήθελα να σας μεταφέρω. Ναι, ήταν πολύ ωραία και συγκινησιακά αυτά που μας είπατε. Η Γιούτα Χάου και μετά ο Βιτόριο. Ähm, Ευχαριστώ πολύ. Προστασία του εδάφους. Όπως είπε και ο Καλχάιντς Φλόρεντς, το 2006 Εφτά τότε συζητούσαμε και όποιος έχει παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση λέει ρε γαμώτο πάλι τα ίδια. Αλλά θα σας πω τι έγινε. Εγώ έλαβα από την Ένωση Γερμανών Αγροτών ε, αυτό το φύλλο εδώ πέρα, δύο σελίδες που έχει πραγματικά πολύ σημαντικές ε, πληροφορίες. Δεν ξέρω αν ρίξατε καμία ματιά. Είναι τα ίδια επιχειρήματα πριν από 5-6 χρόνια. Δεν έχουν μάθει τίποτα. Τα ίδια αντανακλαστικά. Δηλαδή όλα αυτά μακριά από μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ταυτόχρονα επαναλαμβάνουν τις κατηγορίες τους κατά της πρότασης οδηγίας ε, της Κομισιόν. Πουθενά, πουθενά δεν λένε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση είχε κάνει μια θαυμάσια πρόταση. Που την έκανε σαλάτα μετά η Κομισιόν και την ανέτρεψε εντελώς. παρά το ότι είχαμε διακομματική συμφωνία. Αυτό σημαίνει πως αυτό το οποίο μας λέει η Ένωση Γερμανών Αγροτών ε, εν ώψη της ε, συζήτησης αυτής και πως πρέπει να πούμε τη θέση τους ε, το έκανε ο Καλ φτάνει αυτό έτσι το να το λέμε πληροφορία αυτό δεν είναι δυνατόν. Αυτά είναι παραπλανητικά που γράφουν εδώ πέρα. Και ούτω ή άλλω δεν μιλάω πια με κανέναν που δεν αναγνωρίζει πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι νομοθέτης. Und wir haben... Και όχι κομισιόν. Περάσαμε μια πρώτη ανάγνωση επιτέλους. Και επιτέλους Κάποια στιγμή πρέπει να κάνει κάτι το Συμβούλιο για να καταλήξει σε μια κοινή θέση. Για να ε, μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Κατόπιν να πω κάτι στην Κομισιόν. Αν άκουσα σωστά, γιατί δεν ξέρω γιατί γλώσσα μιλάτε. Ε, δεν κατάλαβα τι λέγατε, αλλά άκουγα τα γερμανικά. <laughs> αλλά ε, άκουσα στα γερμανικά πως υπάρχουν προβλήματα με τα δεδομένα. Ε, και τι κάνετε τόσο καιρό. Δηλαδή, πληρώνουμε GMES, έχουμε υπηρεσία ολόκληρη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και από ό,τι κατάλαβα, μια χαρά είναι εκεί πέρα, πολύ καλή δουλειά έχουν κάνει, πάρα πολλές πληροφορίες. Τι σας λείπει δηλαδή από την Κομισιόν, τι πληροφορίες σας λείπουνε. Δεν καταλαβαίνω. Και τι πληρώνουμε εμείς. Σας ευχαριστούμε Γιούτα. Το λόγο έχει ο Βιτόριο Πρόντι, ο οποίος ήταν εισηγητή για τη θεματική στρατηγική τότε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ έχω ανοιχτούς λογαριασμούς με το έδαφος. Όπως είπε και η Γιούτα Χάουγκ, Κάναμε μια καλή δουλειά. Όλοι μαζί. Πρέπει να το πούμε. Και αυτή η δουλειά που κάναμε ισχύει ακόμα. Και μάλιστα έχουμε όλα τα στοιχεία σε ό,τι αφορά το ρόλο του εδάφους στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Άρα, προφανώς το έδαφος είναι ένα σταθερός πόρος, αλλά και σε ό,τι αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου, αλλά και σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι το έδαφος είναι ένα σπάνιο αγαθό, σπάνιος πόρος, Προφανώς, αν τα λάβουμε αυτά υπόψη, προφανώς θα πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη για να ευαισθητοποιηθούν ως προς τον προορισμό του εδάφους. Έχουμε ένα πόρο ο οποίος συρρυκνώνεται. Ε, γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Θα πρέπει να τον κρατήσουμε σε ένα επίπεδο αποτελεσματικότητας, ώστε να τον υψηλότερο. Το έδαφος ε, αποθηκεύει δυο φορές το... Όχι. Περιλαμβάνει ε, διπλάσια ποσότητα άνθρακα από ό,τι ε, έχουμε στην ατμόσφαιρα. Επίσης έχουμε το διοξίδιο του αζότου. Δεσμεύεται Είναι ένα πρόβλημα που μας ενδιαφέρει όλους. Φυσικά θα σεβαστούμε τις θέσεις των κρατών μελών. Φυσικά κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του έδαφους είναι δική του αρμοδιότητα. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, εμείς δώσαμε μάχη για το GMES, την παρακολούθηση από δορυφόρο. Γι' αυτό το φτιάξαμε, για να έχουμε δεδομένα δηλαδή για το έδαφος, για την υγρασία, την κατάσταση των φυτών, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και με μία υποσημείωση Έχουμε όλα τα στοιχεία, έχουμε όλα τα εργαλεία στη διάθεσή μας για να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση του εδάφους. Πρέπει να συνεχίσουμε την ε, μάχη λοιπόν. είναι μια απαραίτητη υποδομή αυτή, το GMES, για την πολιτική μας για το έδαφος και για την πολιτική καταπολέμηση στα αέρια των αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, καταλαβαίνω τα επιχειρήματα για την ε, βελτίωση των μολυσμένων εδαφών. Αν είναι είδος ε, που σπανίζει το έδαφος, όλοι θα πρέπει να συμφωνούμε ότι πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε να βελτιώσουμε το έδαφος, να καθαρίσουμε ε, το μολυσμένο έδαφος, να το κάνουμε πάλι παραγωγικό. Είχαμε αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Και εκεί συζητήσαμε το πώς το έδαφος μπορεί να γίνει ένα αγαθό το οποίο θα το συντηρούμε συνέχεια. Το νερό το οποίο προέρχεται από τη βροχή θα πρέπει να διατηρείται όσο να το περισσότερο, εκεί που πέφτει, για να τροφοδοτήσει τον υδροφόρο ορίζοντα. Επίσης, έχουμε από τη μία τα εδάφη στις αστικές περιοχές. Πρέπει να έχουμε αντιστάθμισμα σε αυτά τα εδάφη στις αστικές περιοχές. Ε, για να μην ε, ε, πάθει καθίζηση το έδαφος, θα πρέπει να υπάρξει έγχυση βρόχινου νερού εκεί, να μείνει εκεί το νερό, να τροφοδοτήσει τον υδροφορορίζοντα. Εγώ είδα και πρόσφατα στοιχεία. Η πόλη της Τζακάρτας έχει κάτσει δέκα φορές περισσότερο από το επίπεδο ανύψωσης, των θαλάσσιων υδάτων. Βλέπετε πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό ειδικά σε μια πόλη όπως η Βενετία. Όλα στο ίδιο καταλήγουν. Όλες οι πολιτικές καταλήγουν πού? Στο έδαφος. Πρέπει να κρατήσουμε το έδαφος στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ούτως ώστε να συνεισφέρει στο καλό και την ευμερία όλων. Πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι δεν υπάρχει καμιά πίεση εδώ πέρα, δεν αναμειγνιόμαστε στις πολιτικές τους. Απλώς υπάρχουν κάποια θέματα που είναι γενικά, που μας ενδιαφέρουν όλες. Ξεκινάμε από την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Να σας υπενθυμίσω τις καταστροφές της Γένοβας και άλλων περιοχών κοντά στη Γένοβα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με μια έλλειψη συντήρησης του εδάφους. Το θέμα είναι όλες αυτές τις γνώσεις να τις ρίξουμε σε αυτό το έγγραφο. Ε, Ούτως ώστε να φτάσουμε σε κάποια πράγματα που τα συμμεριζόμαστε όλοι, όλα τα κράτη-μέλη για το έδαφος, που είναι ένας πόρος στον οποίο πρέπει να επενδύσουμε. Ωραία, βλέπει κανείς την ε, την γνώση και την πείρα που έχετε για το θέμα αυτό. Πόσο καλά ο Βιτόριο γνωρίζει τα θέματα αυτά για το κλίμα και τα εδάφη. Η κυρία Μπελία έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν ήμουν παρούσα το 2006 όταν γινόντουσαν οι συζητήσεις για το σχέδιο οδηγίας για τα εδάφη. Αλλά το 2008 ήμουνα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στα πλαίσια της λεγόμενης Γκρενέλ του Περιβάλλοντος, τις ε, λαϊκές αυτές συνελεύσεις που είχαν λάβει χώρα για τα θέματα αυτά και είδα την επιστροφή του Υπουργού Περιβάλλοντος που είχε πει ότι είχε αντιταχθεί στην ψήφιση της οδηγίας για τα εδάφη και μάθαμε μετά ότι η Γαλλία είχε κρατήσει θέση αποχής. Ναι, καλά, δεν καταψήφισε, αλλά τουλάχιστον έπαιξε κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της ε, ε, μειοψηφίας ανάσχεσης. Ελπίζω λοιπόν ότι σε μερικές εβδομάδες η Γαλλία θα, και φυσικά αυτό εξαρτάται και από τα εκλογικά αποτελέσματα, η Γαλλία θα παίξει και πάλι το ρόλο του κινητήριου, της κινητήριας δύναμης μέσα στα θέματα αυτά και θα τονίσει σε επίπεδο πολιτικό μαζί με τα θέματα της ατμόσφαιρας και του ύδατος να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα εδάφη. Εγώ δεν έχω πάρει τα τελευταία στοιχεία του, από το λόμπι των Γερμανών γεωργών αλλά προσπαθούν να καταλάβουν από πού προέρχεται αυτή η μειοψηφία ανάσχεση. Νομίζω ότι πέραν των ε, στοιχείων που θα πρέπει να κατανοήσουμε που επηρεάζουν τους γεωργούς, νομίζω ότι αυτή η οδηγία έχει ουσιαστικά χρησιμοποιηθεί ως όμοιρος για άλλους στόχους. Οι γεωργοί σε ένα τμήμα της Γερμανίας θεωρούν ότι υπάρχει μια μείωση τη ε, κυριαρχικότητό του ότι χάνουν τα δικαιώματά του, Για αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το έδαφος. Αν δούμε σήμερα ποιε είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολιτικό επίπεδο, για το θέμα αυτό και σε άλλα θέματα θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Εγώ δυσκολεύτηκα να κατανοήσω τα επιχειρήματα σε σχέση με το έδαφος και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορούμε να ρίξουμε το φταίξιμο στα κράτη-μέλη και στους άλλους φορείς για την ανεπάρκεια της εφαρμογής των κανονισμών και των οδηγιών για την... στην Κομισιόν επειδή δεν άσκησε πίεση στα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό η δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου που περιλαμβάνει όλους τους κανόνες της διάφορες κατατομής πολιτικές, είτε πρόκειται για την κλιματική αλλαγή, για την γεωργία, για την αστικοποίηση και όλα αυτά, κατά πόσο συγκροτούν μια συνολική πολιτική για την προστασία των εδαφών μας σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής αν όλα αυτά με το να έχουμε ένα γενικό πλαίσιο θα οδηγήσουν σε επιβράδυνση της πορείας ή δημιουργία προβλημάτων είναι ευκαιρία λοιπόν να προσπαθήσουμε να ξαναβρούμε περισσότερη συνεκτικότητα σε ένα συνολικό πλαίσιο μέσα σε μια πολιτική περιβάλλοντος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ενεργειακά, την κλιματική αλλαγή και να υλοποιήσουμε όλες τις δεσμεύσεις που έχει λάβει υπόψη της και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την βιοπικιλότητα και να καταλήξουμε έτσι σε μια ευρύτερη οδηγία που να έχει ένα ευρύτερο πολιτικό υπόβαθρο όπως έγινε και στην περίπτωση της οδηγίας για την ποιότητα των υδάτων με το να έχουμε στόχους, με το να έχουμε λοιπόν μια διαδικασία η οποία στη συνέχεια θα θέσει ανάγλυφα τα διακυβεύματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των εδαφών. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε λοιπόν ένα πιο πολιτικό διάλογο και σε εθνικό επίπεδο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το έδαφος και τις οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Κλείνω με την εξή παρατήρηση. Εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τις προσπάθειές της. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πρόκειται για μια συζήτηση, βέβαια είναι μικρή η πλειοψήφια που την υποστηρίζει. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την συζήτηση για το 7ο πρόγραμμα του περιβάλλοντος με συγητή το Γιώ Λάινεν ψήφισε αυτό το πλαίσιο για το, τα εδάφη. Φαίνεται ότι είναι σταθερή αυτή η μειοψηφία, αλλά ήταν μια μικρή πλειοψηφία τεσσάρων ψήφων συνεχίζεται η συζήτηση, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχει επιτέλους μια πλειοψηφία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ελπίζω ότι θα μπορέσει να συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Κομισιόν και ο καθένας με το δικό του τρόπο θα πρέπει να ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη ώστε μέχρι το τέλος της θητείας μας να έχουμε επιτέλους αυτή την οδηγία πλαίσιο για τα εδάφη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα η Κομισιόν. Αν θέλει, μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις και μετά τελειώνει η συζήτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τον κύριο Φλόρεντς που ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση με τον τρόπο αυτό. Και να ευχαριστήσω και όλους τους συμμετέχοντες. Θα απαντήσω σε όλες τις παρεμβάσεις μία προς μία. Άκουσα στα πρώτα σχόλια ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της επικουρικότητας και υπέρ της καλύτερης επιτήρησης από πλευράς της Κομισιόν. Όσον αφορά την επικουρικότητα, τα ακούσαμε και από εδώ, η πρόταση της Κομισιόν που είναι και ε, οποιαδήποτε άλλη τροποποίησή της θα αντιμετωπίσει μόνο την διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν σκοπεύει On μπει σε ζητήματα επικουρικότητας και επ' αυτού νομίζω πως το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, οι Γερμανοί αγρότες, όλοι ε, μπορούν να είναι ήσυχοι. Για την εφαρμογή. Εφαρμογή θα ήθελα να πω. Πως είναι πρώτα απ' όλα ευθύνη των κρατών μελών πρέπει τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν την σωστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Και ως έναν βαθμό η Κομισιόν ως θεματοφύλακας της συνθήκης παρεμβαίνει και πρέπει να παρέμβει όταν μιλάμε για μέτρα ελέγχου παρακολούθησης ε, τα οποία δεν λαμβάνονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Δεν γνωρίζω λοιπόν να έχουν γίνει αιτήματα προς την Κομισιόν τα οποία να μην ικανοποίησε. Για τα δεδομένα, τη δεύτερη ερώτηση. Για τα σχόλια GMES, that we have paid for GMES and that they... Ότι δεν υπήρχαν δεδομένα από το GMES και να πάμε να τα πάρουμε από εκεί. Μα το θέμα είναι ποιος έκανε τα αυγό, ποιος έκανε πρώτο το αυγό ή το αυγό την κοτά. Data will never be made available to the Commission. And for this reason, this is one more... Και αυτός είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία πλαίσιο σε αυτό το τομέα. Τα εθνικά δεδομένα μόνο δεν είναι συγκρίσιμα. Κάποια είναι πολύ καλά, πολύ αναλυτικά, κάποια λιγότερο. Δεν είναι όμως συγκρίσιμα. Όσον αφορά το αίτημα ότι η Κομισιόν πρέπει να εξετάσει την οδηγία που το βάλαμε πριν από λίγα έτη και την οποία εξέφρασε η Κομισιόν ε, και βεβαίως ευχαριστούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Βιτόριο Πρόντι για την πρώτη του ανάγνωση και ευχαριστούμε ακριβώ για το ότι υπάρχει μια θέση του Κοινοβουλίου. Εμείς είμαστε έτοιμοι μόλις δούμε την δυνατότητα να ξανατεθεί το ζήτημα. Βεβαίως θα εξετάσουμε όλες τις ε, εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα εν μεταξύ. Δεν θα ήταν σωστό να βάλουμε στοιχεία πριν από 5 ή 6 έτη. Αλλά πρέπει να βρούμε την κατάλληλη στιγμή. In the meantime, I can only say that Εν τω μεταξύ έχουμε ενθαρρύνσεις από διάφορες ε, πλευρές και ακόμα ε, και τις λιγότερο θετικές ε, πλευρές από λίγα χρόνια. Σε λίγε μέρες ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα σχόλια τα οποία θα έχουμε συλλέξει περισσότερε πληροφορίε θα υπάρξουν κάποια γεγονότα τα οποία θα λάβουν χώρα μέσα στο πλαίσιο των πραγματικών διαπραγματεύσεων σε σχέση με τα εδάφια, όπου θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του εδάφου σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά το θέμα των εδαφών δεν είναι μόνο ένα παγκόσμιο θέμα. Είναι ένα θέμα και ευρωπαϊκό. το γεγονός ότι τα εδάφη στεγανοποιούνται. Όλα αυτά είναι θέματα που οποία μας απασχολούν. Σας ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρος στην Κομισιόν. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους οι οποίοι έλαβαν μέρος στην συζήτηση. Πιστεύω ότι ήταν όλα αυτά πάρα πολύ χρήσιμα και είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά δεν έχει φτάσει στο τέλος του προβληματισμού. Ε, υπάρχουν πολλά ακόμα ζητήματα τα οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο στις 7 Μαΐου από τις 3 ως 6.30 θα συνεδριάσουμε και την επόμενη στις 8 Μαΐου το πρωί. Όλα αυτά θα γίνουν στο διαδίκτυο. Επίσης θα μπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο με web streaming και στην ε, βιδεοθήκη του Κοινοβουλίου. Όλα αυτά τα συναρπαστικά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε λοιπόν. Και σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα και καλές γιορτές.